Alors, chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà. Euh, να ξεκινήσουμε σήμερα το πρωί. Στην συνεδρία της Επιτροπής μας υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο σχέδιο μερίσιας διάταξη. Στις 10 και 4 θα συζητήσουμε τον κατάλογο των τρίτων χωρών, των οποίων οι υπήκοοι υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κατών μελών και τρίτων χωρών, οι επίκο των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή του ψηφοπαίδου τη κυρία Φαγιών. Και ξεκινάμε τώρα με την κατάσταση έκτακτη ανάγκη στη Γαλλία και το κατά πόσον ε, αυτό συμμορφούνται με το πρωτογενέ και δευτερογενέ δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγα λόγια, το ιστορικό αυτή τη νομοθεσία, λόγω των επιθέσεων μεγάλη κλίμακα στι 13 Νοεμβρίου του περασμένου έτου, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν νόμο επί της Η παράταση της κατάστασης αυτής για τρεις μήνες από τις 20 Νοεμβρίου του 2015 εγκρίθηκε από το Γαλλικό Κοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2015 και στις 19 Φεβρουαρίου 2016 για μια νέα τριμήνη περίοδο και για άλλους ε, δύο μήνες στις 20 του περασμένου μήνα. Η έκτακτη ανάγκη ορίζεται στη γαλλική νομοθεσία με τη θέσπιση κάποιων μέτρων που μπορούν να λάβουν οι διοικητικές αρχές και κάποια από τα μέτρα αυτά μπορεί να οδηγήσουν στις, σε εξαίρεση από τις υποχρεώσεις διαφύλαξης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Μετά τις 24 Νοεμβρίου του 2015, 19 ε, Φεβρουαρίου και 25 Μαΐου του 2016, οι Γαλλικές Αρχές ενωμέρωσαν τις αρχές του Συμβουλίου ότι θα χρησιμοποιήσουν την παρέκκληση του άρθρου 15 βάσει της απόφασης και βάσει της απόφασης των συντονιστών θα ακούσουμε τον κύριο Πιέρ Σελάλ έκτακτο πρέσβη παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνιμο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα εκτεσανάκη ανάγκη στη Γαλλία και την ε, συμβατότητα των μέτρων αυτών και το κατά πόσο είναι συμβατά από την Ευρωπαϊκή Πρωτογενή και Δευτερογενή Νομοθεσία. Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τα συλληπιτήριά μας ε, μετά την ε, ε, δολοφονία του αστυνομικού και τη συζύγου του στις 13 Ιουνίου, προχθές. Θα έχουμε πρώτα μια σύντομη παρουσίαση από τον κύριο Σελάλ και μετά θα προχωρήσουμε ως συνήθως σε ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Σελάλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Είναι προνόμιο και τιμή να μπορώ να μιλήσω ενώπιόν σας και να απαντήσω στις ερωτήσεις και σε οποιαδήποτε αιτήματα έχετε για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Γαλλία. Θα ήθελα επίσης να σας ε, ευχαριστήσω για τα συλληπιτήρια που εκφράσατε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, επίθεση που έγινε πριν από τρεις ημέρες ε, στη Γαλλία. Τι είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το περιγράψατε κυρία Πρόεδρε. Είναι μια ειδική κατάσταση που περιγράφεται από το δίκαιο και χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τον ε, νόμο του 1955 από μία κατάσταση έκτακτου κινδύνου που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα είτε λόγω φυσικών καταστροφών είτε λόγω δημοσίου κινδύνου. Πρόκειται λοιπόν για μία πολύ αυστηρή νομική περιγραφή του κινδύνου αυτού. Δεν είναι ένα πολιτικό ζητούμενο. Είναι μια νομική κατάσταση σύμφωνα με την οποία ε, οι διοικητικές αρχές έχουν το δικαίωμα να έχουν συγκεκριμένα προπ προνόμια σε όλο το έδαφος της χώρας. Είναι μια λογική πρόληψη ε, στην ουσία που έχει εμπνεύσει αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουμε να προλάβουμε πιο ε, δύσκολα προβλήματα που προκύπτουν σε τέτοιες εξαιρετικές ε, καταστάσεις. Αμέσως μετά λοιπόν τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου κηρύχθηκε η κατάσταση του έκτακτης ανάγκης και μετά ε, παρατάθηκε για τρεις μήνες, τον Φλεβάρι άλλες, άλλους τρεις μήνες ε, και στις 20 Μαΐου πάλι ε, δόθηκε άλλη μία παράταση. Άρα σήμερα ισχύει ακόμα. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα, κάποια μέτρα που υιοθετήθηκαν και σύμφωνα με την ομοθεσία και σύμφωνα και με τους δικαστές αυτά είναι απαραίτητα και αναλογικά. Δεν υπάρχει ε, λοιπόν τώρα το δικαίωμα διαμαρτυρίας ε, και διαδηλώσεων γιατί πρέπει να αποφύγουμε τη συγκέντρωση ανθρώπων διότι μπορούν να αποτελούν έναν δυνητικό στόχο για κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις ε, και για να αποφύγουμε κάποια παρεκτροπή που θα μπορούσε να θέσει υπό την ασφάλεια. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της διάσκεψης για το κλίμα που έγινε το Δεκέμβρη ε, στο Παρίσι ε, αποφασίστηκε αυτή η απαγόρευση των διαδηλώσεων. Όπως ε, παρατηρήσατε, βέβαια, η κοινωνική κατάσταση στη χώρα μου αυτή τη στιγμή είναι διαφορετική. Υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Δεν είναι λοιπόν γενική και απόλυτη αυτή η απαγόρευση οι διοικητικές αρχές ε, στην ουσία προσαρμόζουν ε, αυτά τα μέτρα απαγόρευσης. Επίσης ε, μιλάμε για διοικητικές έρευνες όταν υπάρχει αυτή η ανάγκη και αυτό είναι εάν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν λάβει μέρος σε δράσεις που θέτουν σε κίνητο τη δημοκρατία. Μιλάμε λοιπόν για διοικητικέ έρευνες και βάσει ε, του απολογισμού που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες, ε, περίπου στις 15 Μαΐου, Είχαμε 3.427 τέτοιες έρευνες που έγιναν ε, κατά κύριο λόγο την πρώτη περίοδο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δηλαδή μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου. Από τις 26 ε, Φεβρουαρίου μέχρι τις 9 ε, Μαΐου είχαμε 145 τέτοιες έρευνες, διότι φυσικά τα περισσότερα είχαν γίνει στην πρώτη περίοδο. σύμφωνα με τα αποτελέσματα 750 όπλα μπόρεσαν να ε, εξουδετερωθούν βάσει αυτών των ερευνών. Το πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα ήταν ε, η ε, ενημέρωση που στην ουσία επιτεύχθηκε και μπόρεσε να μας κάνει να μην έχουμε πλέον αμφιβολίες, να ενημερώσουμε τους φακέλους και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι πάνω από τις μισές έρευνες έχουν να κάνουν με άτομα που ήταν ήδη ε, στους φακέλους της αστυνομίας. Επίσης υπήρξε μία άλλη ε, έρευνα ε, δικαστική. Οι 59 από τις ε, διοικητικές έρευνες οδήγησαν σε δικαστική έρευνα, πρώτον λόγω της, νοσοκο... της νομοθεσίας για τα όπλα, δεύτερον λόγω της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Και αυτές οι έρευνες μπόρεσαν να μας επιτρέψουν να δούμε την κατάσταση, να δούμε πόσο διαπερατή είναι η ε, εγκληματικότητα. Υπάρχει σχέση μεταξύ της τρομοκρατίας, ε, του εμπορίου όπλων και ε, των ναρκωτικών. Οι κρατήσεις κατοίκων με 268 διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει το Φλεβάρι οδήγησαν σε τρεις κρατήσεις κατοίκων ε, αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μετά από πρόσφατες αποφάσεις. Τέλος, να σας επισημάνω ότι ενώ η κατάσταση εκτακτής ανάγκης δίνει τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να περιορίσουν την ελευθερία συγκέντρωσης, μόνο ε, ένας τόπος άσκησης θρησκευτικών κατοικούντων ε, έπαψε τη λειτουργία του. Αυτή είναι η κατάσταση. Βεβαίω, εσεί ανησυχείτε για να ξέρετε και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο όλων αυτών των μέτρων και το βουλευτικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο. που οδήγησε στην άσκηση αυτών των μέτρων. Υπάρχει ένα σημείο για το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Η κατάσταση εκτεκτή ανάγκης δεν σημαίνει ότι έχουμε παραμερίσει το κράτος δικαίου. Τα μέτρα που προβλέπονται ε, υπόκεινται σε μια σειρά από εγγύησεις και ελέγχους. Οι εγγυήσει ε, σημαίνουν ότι 20 Νοεμβρίου του 2015 με την απόφαση που ελήφθη έχουμε τουλάχιστον εφαρμογή δύο νόμων που έχουν προβλεφθεί το 1965 όπως η κατοίκον κράτηση. Άλλαξε το πεδίο εφαρμογής του νόμου για να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα της απειλής, να υπάρχει περιορισμός στο χώρο και το χρόνο της άσκησης των μέτρων και να εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα για τις ε, κατοίκων έρευνες ε, διοικητικού τύπου χρειάζεται η εντολή του εισαγγελέα, η παρουσία αστυνομικών αρχών για να προχωρήσουν σε δίμευση κατάσχεση και η διαρκής ε, μετάδοση πληροφοριών στον εισαγγελέα, καθώς και η πρόβλεψη μέτρων για ορισμένους φορείς όπως βουλευτές, δικηγόροι, οι οποίοι ε, δεν μπορούν να είναι σε καμία περίπτωση αντικείμενο κατοίκου κράτηση. Επίσης πλαισίωση από το δικαστή. Ο συνταγματικό δικαστή σημαίνει ότι το Συμβούλιο επικρατεία που πόκειται στη γαλλική μας δικαιοδοσία όπως ενέκρινε με την απόφασή του τη 20 Δεκεμβρίου του 2015 ενέκρινε τη συνταγματικότητα των ε, μέτρων αυτών της κατοίκων κράτησης και, και το, την άσκησή τους. Η απόφαση του δικαστή που ήταν ε, και η προϋπόθεση για να εγκριθεί συνταγματικότητα και άσκηση των μέτρων αυτών ε, αποφάσισε και κατέληξε στο πόρισμα ότι είναι αναλογικά και δικαιολογημένα τα μέτρα αυτά. Έτσι ε, προβλέπει η γαλλική νομοθεσία, όπως συγκρίνει και το Συμβούλιο Επικρατείας από το 1930. Για τις διοικητικές κρατήσεις κατοίκων, το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφασή του του Φεβρουαρίου του 2016 διευκρίνησε ότι οι διοικητικές αρχές δεν μπορούν να αντιγράφουν τις ε, ε, αποφάσεις χωρίς την, απόφαση, την πρώτη απόφαση ενός διοικητικού δικαστή, προτού αποφασιστεί ε, η διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν η διαδικασία να εγκρίνεται και να πλησιώνεται και η υλοποίησή της. Στην ε, Γαλλία διοικητική διαδικασία μπορεί να είναι και το Συμβούλιο Επικρατεία, όπω γίνεται με τα ασφαλιστικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα περιορισμού τη ελευθερία, ε, που μπορεί να προβλέψουν την ε, στέρηση ελευθερία σε περίπτωση που υπάρχει δια... πράξη άδικη παράνομη και να στερηθούν και παραβίαση θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει λοιπόν με τα πρώτα εκτελεστικά μέτρα. Πρώτος απολογισμός έγινε στα τέλη Απριλίου του 2016 από το Συμβούλιο Επικρατείας που κατέληξε στον αριθμό ότι για το 1 τρίτο, το 1 τρίτο των αποφάσεων για άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατεπηγόντως, 38 από 111 έχουν ε, ε, αμφισβητηθεί μπροστά στον ε, δικαστή που κρίνει την απόφαση άσκηση ασφαλιστικών μέτρων. Είτε τι ε, απορρίπτει, είτε τι ανακαλεί, ε, τι καταργεί. Αυτό δείχνει ότι ο έλεγχο του διοικητικού δικαστή για τα μέτρα που λαμβάνονται ασκείται πραγματικά και πολύ συχνά οδηγεί στην αναστολή, την ακύρωση ή την ε, μη εφαρμογή, την κατάργηση των μέτρων που έχουν αναλυφθεί. Η κατάσταση λοιπόν έκτακτη ανάγκη και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε αυτό το πλαίσιο δεν σημαίνει ότι έχουμε σταματήσει να, να σεβόμαστε το κράτο δικαίου και να υποκείμεθα στου κανόνε του. Απλώ οι διάφορε υπηρεσίε και αρχέ έχουν ιδιαίτερο έλεγχο δικαστικό σε σχέση με πριν ο νομοθετικός έλεγχος, ο έλεγχος των δικαστών και βουλευτικός έλεγχος επίσης. Ο νόμος της 20 Νοεμβρίου 2015 προβλέπει έλεγχο ε, βουλευτικό κοινοβουλευτικό α, ε, της άσκησης των μέτρων αυτών, η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία ε, ενημερώνονται αμελητή για την λήψη μέτρων από την κυβέρνηση, δίνοντας περαιτέρω πληροφορίες στα πλαίσια του ελέγχου και της αξιολόγησης των μέτρων αυτών. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η νομική επιτροπή της Εθνοσυλλέλευσης και της Γερουσίας ε, λαμβάνουν ε, συστηματικά αριθμητικά δεδομένα από την κυβέρνηση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ε, μπορούν να ανταλλάξουν επιστολές με το Υπουργείο Εσωτερικών. 66 ανταλλάχθηκαν ως τώρα. Ε, διενεργούν ακροάσεις σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών, Άμυνας, σε επίπεδο Δημοτικών Αρχών και ο βουλευτικό έλεγχο υπήρξε πραγματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη περίοδου. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, το είπατε και στην εισηγήσή σα, κυρία μου, τα μέλη τη Επιτροπή σα αναρωτιόνται κατά πόσον το, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Γαλλία συνάδει και με τις διεθνεί μα υποχρεώσει, συγκεκριμένα με τη σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να ασκήσει, να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις που υπάρχουν και στο Διεθνές Σύμβολο για τις πολιτικές ε, και αστικές ελευθερίες, του άρθρο 4, και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρθρο 15, που προβλέπει παρέκκληση όταν ένα κράτος για συγκεκριμένους λόγους μπορεί να ε, αναστείλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την άσκηση προσωπικών και θεμελιωδών ελευθεριών σε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Ακριβώς αυτό δηλαδή που ε, ε έχει οδηγήσει στην πρόβλεψη η κατάσταση της ανάγκης στη χώρα μου. Το σημείο στο οποίο θα επιμείνω ακόμη μια φορά είναι ότι αυτή η παρέκκληση και η δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει από το πεδίο της σύμβασης. Πρόκειται για νομικά εργαλεία, για νομικέ δυνατότητε που προβλέπονται από αυτά τα δύο μέσα και σημαίνει ότι με συγκεκριμένε διαδικασίε, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, λόγω των έκτακτων περιστάσεων, όπως προβλέπουν οι διεθνείς συμφωνίες, μπορεί να ισχύσουν αυτές οι εξαιρέσει. Αυτό προβλέπεται και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της ε, εφαρμογή αυτών των δύο νομικών εργαλείων. Έτσι λοιπόν, από αρκετού μήνε έχουμε συστηματικέ ε, συνεννοήσει με του ειδικού επετετραμένου του ΟΗΕ και ιδίω το υπευθύνου τη Επιτροπή τη Βενετία. Επιτροπή τη Βενετία, η οποία νομίζω επισκέφθηκε την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Εσωτερικών και ο υπεύθυνό μα για τι ευρωπαϊκέ υποθέσει πήγαν στο Στρασβούργο για να ενημερώσουν τον ε, Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Επίσης, ε, το Φεβρουάριο στη Γενέβη παρουσιαστήκαμε και στην Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για να εξηγήσουμε τι συμβαίνει με την κατάσταση εκτεκτής ανάγκης στην ε, Γαλλία, εξηγώντα τα έκτακτα μέτρα που αναλήφθησαν και ε, εξηγώντα ότι μα απασχολεί η ασφάλεια των πολιτών και η άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών ούτω ή άλλω. Δίνουμε μεγάλη προσοχή σε αυτά στη Γαλλία. Τελευταία παρατήρηση διερωτηθήκατε ποιος είναι ο λόγος παράτασης επανειλημμένος της ισχύω κατάστασης εκπαιδευτικής ανάγκης και για τελευταία φορά πριν από λίγες εβδομάδες μόλις. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας είπε ξεκάθαρα ότι η κατάσταση εκπαιδευτικής ανάγκης δεν πρόκειται να διαρκέσει Όμως ευθύνη του είναι να βεβαιωθεί για την ασφάλεια των πολιτών όταν η απειλή και ο κίνδυνος παραμένουν ε, παρόντες. Η Γαλλία νομίζω ότι συνεχίζει να αποτελεί ένα στόχο, ε, κατεξοχήν στόχο, για τις τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδίω του τσιχαντιστές, κυρίως για τις επιθέσεις του, κατά, για τις επιθέ... λόγω των επιθέσεων της, κατά των τζιχαντιστών, του ISIS, στο... στην, στην περιοχή του Μάλι, τη Ιράκ και τη Συρίας. Η χώρα μας εκπροσωπεί κάποιες θεμελιώδεις αξίες που είναι παράδοσή μας εδώ και αιώνες και γιατί ακριβώ μας αποτροπιάζουν οι τρομοκράτες και οι τζιχαντιστές. Θεωρούμε λοιπόν ότι η απειλή παραμένει υψηλή και παρούσα και η αποτροπή μεγάλης επίθεσης τον Μάρτιο, επίθεση η οποία προβλέπεται να είναι μεγάλης κλίμακας, είναι μια απόδειξη. Εδώ και δύο χρόνια 12 επιθέσεις έχουν αποτραπεί και αναφερθήκατε σε νέα επίθεση που έγινε μόλις πριν από τρεις μέρες. Δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους δύο αστυνομικοί, δολοφονήθηκαν απλώς γιατί ήταν αστυνομικοί. Ζούμε σε καταστάσεις που πραγματικά ε, επιβάλλουν το να είμαστε διπλά προσεκτικοί, όπως ε, η διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, όπου συμμετέχουν 2,5 εκατομμύρια φίλαθλοι και θεατές, η έλευση στη Γαλλία 8 εκατομμυρίων ανθρώπων ε, με τον ένα τον άλλο τρόπο ε, δικαιολογούν την εξαιρετική προσοχή που πρέπει να δώσουμε για τις αθλητικές αυτές εκδηλώσεις και τη διοργάνωσή τους. Βεβαίως, μεγάλη προσπάθεια έγινε και ως προς τα μέτρα προστασίας του φύλαθλου κοινού και για να σας πω απλώς έναν αριθμό, 110.000 αστυνομικοί έχουν αναλάβει δράση στην επικράτειά μας, χωροφύλακες, αστυνομικοί και ε, άλλοι πράκτορες, οι οποίοι θεωρούν ότι η ε, αιμονή του κινδύνου αυτού δικαιολογεί την παρουσία τους. Η διοργάνωση Ήδη είδαμε τα περιστατικά μεταξύ πολιτών ε, λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Γαλλία. Ε, σας τα θύμισα και προηγουμένως. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι για τους οποίους για άλλη μια φορά η κατάσταση εκτός ανάγκης συνεχίζει να ισχύει στη Γαλλία, αλλά ε, επιμένω ότι πρόκειται για ένα πλαισιωμένο ε, νομικό σύστημα το οποίο δικαιολογείται, έχει προσαρμοστεί στις συγκεκριμένε ανάγκες και διαρκώ φροντίζει να συνδυάζει την προστασία των ε, προσωπικών ελευθεριών, των θεμελιωδών ελευθεριών, με τις ανάγκες προστασίας της δημόσιας τάξης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη, για αυτή την παρουσίαση που μας δώσατε με πολλές λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσουμε τώρα ακούγοντα ερωτήσει των συναδέλφων. Πρώτα απ' όλα τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο κύριος Έγγελ. Έχω δύο-τρεις σκέψεις που θα ήθελα καταρχήν να μοιραστώ μαζί σας. Θα ήθελα να δω καταρχήν πώς είναι ακριβώς ε, η εφαρμογή, γιατί ε, ξέρετε, όταν μιλάμε για μια κατάσταση επίγουσα ανάγκη, δεν μπορούμε βέβαια να την διονύζουμε και να θεωρήσουμε πως η διάρκεια τη θα είναι αόριστη. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχει αυτό ο κίνδυνο είτε στη Γαλλία είτε αλλού για τον απλό λόγο πως μοιάζει επειδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα τα οποία μεν δεν είναι καινούργια αλλά έχουν εντυπωσιακοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε πως οι ανακριτικές μας διαδικασίες και κανόνες είναι ανεπαρκείς και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για όσους έχουν ε, μαθητεύσει στο γαλλόφωνο δίκαιο η νομοθεσία στο παρελθόν απαγόρευε ρητά τις κατοίκων έρευνες για το θέμα της μοιχείας το οποίο οδηγούσε σε πολύ περίεργες καταστάσεις όπου ο κόσμος έπρεπε να σηκωθεί στις 4.30 ώρα το πρωί έτσι ώστε να είναι κρύο το κρεβάτι τη στιγμή που μπορούσε πια γιατί ήταν πρωί να μπει ο αστυνομικό στο σπίτι για να ελέγξει κατά πόσο είχαμε περίπτωση μοιχείας ή όχι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε το κρεβάτι να μην είναι ζεστό. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό δεν δικαιολογείται. Και αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα, και μιλώ βέβαια και με αστυνομικού και με αστυνομικέ υπηρεσίε ε, και με άλλε υπηρεσίε, πω έχουμε παραβιάσεις για τις οποίες χωρίς τέτοιου είδους ε, κατάσταση επίγουσας ανάγκη θα μπορούσαμε να αλλάξουμε προσέξη και να πούμε πως, για παράδειγμα, οι κατοίκον έρευνες, εάν στις 11.30 ώρα το βράδυ θεωρήσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να μπούμε σε ένα σπίτι να το ψάξουμε, να το κάνουμε. Και να μην χρειάζεται να επικαλεστούμε την κατάσταση επίγουσας ανάγκης για να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι αυτό ε, θα ε, καταπατήσει τα δικαιώματα κάποιου στην οικογενειακή ηρεμία θα είναι μια δυνατότητα της αστυνομία να είναι πιο αποτελεσματική. Για μένα λοιπόν αυτή η κατάσταση επίγουσα ανάγκη, παρόλο που όπως είπατε και εσείς νομικά α, πλαισιώνεται θα πρέπει να περιοριστεί ακριβώ στις περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη και στη Γαλλία είχαμε τις επιθέσεις, τη διάσκεψη των Παρισίων λίγο μετά πάρα πολλοί κόσμος, ε, κίνδυνοι ασφαλής εντάξει Παράταση λοιπόν και όπως είπατε και εσείς Έχουμε το, ε, ε, γαλλικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα του Ευρωπαϊκού του Ποδοσφαίρου, έχουμε το γύρο της Γαλλίας. Άρα λοιπόν πιστεύω πως δεν χρειαζόμαστε κατάσταση επίγουσας ανάγκης, χρειαζόμαστε διαδικασίες οι οποίες να είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους απειλές. Και για να το κλείσω, πέρσι, τέτοια εποχή, εγώ διάβαζα στην εφημερίδα Le Monde πως υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες τζαμιά ή τουλάχιστον 100 τζαμιά ε, ριζοσπαστικοποιημένα στη Γαλλία. Δεν συλλαμβάνονται οι μάμιδες οι οποίοι προσιλητίζουν προς το ριζοσπαστικισμό και δεν τους εκδίδουμε σε άλλη χώρα ή δεν τους διώχνουμε. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε πολλά. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε πει ε, να το αντιμετωπίσουμε χωρίς την κατάσταση πήγουσας ανάγκης γιατί βέβαια έχουμε μια ανεκτικότητα, αλλά ανεχόμαστε φαινόμενα τα οποία μας απειλούν και για τα οποία θα πρέπει να αλλάξουμε τουλάχιστον τη νομική στάση που τηρούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έγκελ Από τους ε, σοσιαλιστέ, σοσιαλιστές η κυρία Τσίπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πολύ αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης στη Γαλλία και ε, των δυνατοτήτων που υπάρχουν βάσει της κατάστασης ε, έκτακτης ανάγκης. Συμφωνώ με τον κύριο Έγγελ ότι όταν υπάρχει κίνδυνος ε, θα πρέπει και θα μπορούμε να έχουμε πιο ευέλικτη χρήση των κανόνων και όταν αυτό έχει επιπτώσεις στην κοινωνία γενικά, καλό θα είναι αυτές οι καταστάσεις να μην διαρκούν πολύ. Ε, όπως γνωρίζετε, ε, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη δύσκολη κατάσταση στη Γαλλία. Όμως υπάρχουν ε, κάποιες συμπληρώματα σε αυτή την νομοθεσία ε, που έχουν να κάνουν με άλλες σκέψεις, ας πούμε για παράδειγμα ε, των μέτρων που έχουν ληφθεί για το Euro, για το γύρο της Γαλλίας, για τις απεργίες, έχουν να κάνουν ε, με την διαφορετική διάρθρωση και στελέχωση της αστυνομίας. Ε, υπάρχουν σκέψεις ε, να εκπαιδευτεί η αστυνομία αλλιώς. Ε, έχει γίνει μια συζήτηση για προληπτικά μέτρα ε, που θα λαμβάνονται εκ των προτέρων ε, και μεσοπρόθεσμα να μπορεί κανείς να άρει αυτό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Επίσης αναφερθήκατε σε κατασχέσεις, είπατε και σε ότι σε 3.427 έρευνες βρέθηκαν όπλα σε πόσους βρέθηκαν σε ε, μία, σε πέντε έρευνες, ε, ήταν μεμονωμένα όπλα. Ε, όλα αυτά είναι σημαντικά. Πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η παράνομη κατοχή όπλων. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποθήκες όπου βρίσκονται αυτά ή μέρη που τα συγκεντρώνουν. Επίσης για τη χρηματοδότηση υπάρχει, όπως είπατε, η σχέση του εμπορίου ναρκωτικών και όπλων με, τον, με την τρομοκρατία. Όμως μέσα στα πλαίσια των ερευνών και των ε, κατασχέσεων αυτών των 750 περιπτώσεων, δηλαδή υπήρχε συγκεκριμένη σχέση και άμεση σύνδεση με αυτό την τρομοκρατία, τα άτομα αυτά συμμετείχαν στις επιθέσεις ή ήταν κυρίως έμποροι ναρκωτικών και όπλων που δεν είχαν σχέση με την τρομοκρατία. Και μια τελευταία ερώτηση αναφέρατε ότι έχουν ξεκινήσει ποικίλε ποινικέ διαδικασίες. Πόσες είναι αυτές, ε, ποια είναι τώρα η, ε, το στάδιο, σε ποια κατάσταση είναι και ε, ποιος, ποια η αιτία, οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατία είναι η κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ. Η ΙΣΙΑΡ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Αλαάου. Πρέπει να σας πω πως αντιμετωπίζουμε συνέχεια καταστάσεις οι οποίοι μας οδηγούν στο να παρατείνουμε αυτές τις καταστάσεις επίγουσας ανάγκης ε, και όντως υπάρχουν οι λόγοι που μας οδηγούν σε αυτό. Όμως η απειλή της ε, ε, των ριζοσπαστών μουσουλμάνων είναι συνεχής. Δεν μπορούμε εμείς λοιπόν να συνεχίζουμε σε ένα καθεστώς επίγουσας ανάγκης, γιατί βέβαια μπορεί να αντιμετωπίζουμε απειλές αλλά ίσως θα έπρεπε να δώσουμε μια άλλη απόκριση με διαφορετικές δράσεις και να εφαρμόσουμε κανόνες οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε ταχείες επεμβάσεις και πιο συγκεκριμένες χωρίς να έχουμε ανάγκη αυτή την κατάσταση ε, σας ανάγκης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρισπέρκ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη που δεχτήκατε να έρθετε να μας κάνετε αυτή την, την παρουσίαση και κυρίως για αυτό το διάλογο που έχουμε, ο οποίος ε, δυστυχώς από πολιτικής άποψης έχει καταστεί όχι τετριμένος, αλλά τουλάχιστον ε, πιθανός και λαμβάνει χώρα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ε, έχουμε ακούσει επανειλημμένως εκπροσώπους κατών μελών, όπου εφαρμόζεται ιδιαίτερη κατάσταση νομική στην ε, περίπτωσή τους όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Δανία και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που δεχθήκατε αυτόν τον διάλογο, αυτή τη συζήτηση που είναι αρκετά ε, δύσκολη και βεβαίω ε, έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη χώρα μα στη Γαλλία. Είναι τολμηρή η απόφαση. Είναι τολμηρέ οι αποφάσει που πρέπει να λάβουμε. Ευχαριστούμε για την πλήρη παρουσίαση, για το νομικό πλαίσιο και τις επιπτώσεις των νομικών αποφάσεων και το πώς η Γαλλία τοποθετείται σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες, τις παρεκκλήσεις, όταν προβλέφθηκαν όλες αυτές οι εξαιρέσεις από τα όσα ισχύουν και ευχαριστώ και για τη σαφήνεια σε σχέση με τα νομοθετικά βήματα που έκανε η χώρα μας, η Γαλλία, ιδίως στο δεύτερο εξάμενο της περασμένης χρονιάς και το πρώτο εξάμενο αυτής της χρονιάς, το 2016, σε σχέση με το νόμο του 2006, του Μαΐου 2016, που μπορεί να προβλέψει καταστάσεις λίγο πιο σταθερές και λιγότερες εξαιρέσεις σε σχέση με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ένα ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που προβλέπεται και έχει και την ε, ανάλογη πλαισίωση, ενώ αρχικά είχε θεωρηθεί κάτι προσωρινό. Έχω λοιπόν αρκετές ανησυχίε Έχω συνείδηση μάλλον ως Γαλλίδα και υπάρχουν πολλοί Γάλλοι από το Κοινοβούλιο για την κατάσταση διαρκούς έντασης των διαρκών ε, συνεννοήσεων που χρειάζονται σήμερα και την ε, κατάσταση μόνιμης απειλής που είναι αρκετά σαφής και συνοδεύεται από μία σειρά αναβρασμού θα έλεγα σε κατάσταση στο επίπεδο των πολιτών με διαδηλώσεις σημαντικές, με διαμαρτυρίες για τα κοινωνικά δικαιώματα. Και για να ολοκληρώσω με αυτά τα προκαταρτικά σχόλια και μετά θα συντομεύσω, θέλω να πω ότι από πλευράς μου θεωρώ ότι η δήλωση για την ε, εφαρμογή της κατάστασης έκπαικτης ανάγκης μετά την γεγονότα της 13ης Νοεμβρίου είναι απόλυτα δικαιολογημένη σε σχέση με τις ε, περιστάσεις. Όμως, ταυτόχρονα, άκουσα με μεγάλη προσοχή. Θα μπορούσατε να είσαστε και καθηγητής ε, δικαίου. Και για να χρησιμοποιήσω την ωραία διατύπωση των νομικών, η ελευθερία είναι κανόνας και τα αστυνομικά μέτρα η εξαίρεση. Αλλά η μεγάλη διάρκεια της εφαρμογής κατάστασης εκτακτής ανάγκης και υπό τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που αναφέρατε καταλήγει να αποδυναμώσει το νομικό ε, σύστημα και την αποτελεσματικότητα της ε, ιδιαίτερης αυτής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ε, η μεγάλη λοιπόν διάρκεια αυτής της κατάστασης, ενώ ο προσωρινός χαρακτήρας της άσκησής του επιτρέπει στο κράτος να ανταποκριθεί σε κάποιες συγκεκριμένε ε, δυσκολίες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι ίδιοι οι Γάλλοι πολίτες δεν συνειδητοποιούν ότι ισχύει καθεστώ έκτακτη ανάγκη. Και η δεύτερη ερώτησή μου, που είναι περισσότερο νομική, είναι ότι ο στόχο αυτή τη κατάσταση έκτακτη ανάγκη είναι να προσπιστεί όχι το κράτο το ίδιο, αλλά το κράτο δικαίου ε, κατεξοχήν η κατάσταση έκτακτη ανάγκη ε, δεν μπορεί να είναι ένα τετελεσμένο γεγονός όπως το κράτο δικαίου και ε, αποδυναμώνονται οι εξαιρετικέ αρμοδιότητες που προσδίδει το καθεστώ αυτό. Τα εξηγήσατε κι εσείς. Ε, οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν επιγόντω, οι αποφάσεις να μην διοργανωθούν διαδηλώσει, να απαγορευτούν. Το είπατε κι εσείς, η φρικτή επίθεση που ζούμε σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά αυτό που έγινε στη Γαλλία πριν από δύο μέρε. Δείχνουν όλα αυτά ότι η αποτελεσματικότητα του καθεστώτο έκτακτη ανάγκη ε, αποδυναμώνεται. Κυρία Γκρισμπέκα, μπορείτε συντομεύετε. Ήθελα λοιπόν να ξέρω τι διαβαθμίσεις μπορεί να υπάρξουν. Ε, δεν είμαστε και σε πολιορκία και πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις απαντήσεις μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Βερζιά, έχετε το λόγο από Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για την νομική αυτή έκθεση ε, που βασίζεται πάρα πολύ, έχει μεγάλη θεμελιώνη την ε, κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει αυτή τη στιγμή ισχύει στη Γαλλία. Συμφωνώ ε, με κάποιες από τις ανησυχίες που έχουν οι πολλοί Γάλλοι για αυτά τα μέτρα. Καταρχάς, ε, είμαστε σε μια κατάσταση κατεξαίρεση που επίσης δικαιολογεί μέτρα κατεξαίρεση. Όμως, ε, ταυτόχρονα, ε, πολλές, πολλά από αυτά παραβιάζουν τις αρχές του κράτους δικαίου, συγκεκριμένα τις ατομικές ελευθερίες που αμφισβητούνται εξ ονόματος αυτής της απαραίτητης ανάγκης. Θα σας πω κάποια περι πράγματα. Έχουμε ένα ε, νόμο το 1955 που ε, εκείνη την εποχή λοιπόν ε, ήταν απαραίτητος γιατί ήταν μια εξαίρεση τότε, αλλά υπήρχαν κάποιες αναταραχές σε λαϊκές συνοικίες. Αυτός ο νόμος τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο και ενισχύθηκε ε, όχι στον πόλεμο της Αλγερίας, αλλά ε, μετά τις ε, ε τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου. Αναρωτιέμαι λοιπόν, έχει δίκιο η Ναταλία που λέει αυτά που λέει, όμως σύμφωνα με τις έρευνες υπάρχει ένα συγκεκριμένος τρόπος που διεξήχθηκαν κάποιες έρευνες και που δεν δικαιολογούνται σε ένα κράτος δικαίου. Επίσης, το να πάει κανείς κατοίκον και να... Ε, ψάχνει να πηγαίνει σε οικολόγους ε, και να λες ε, τι σχέση έχουν με την τρομοκρατία. Ναι, και να τους έχει σε επεκατοίκον κράτηση. Όντως το Μάη έχει γίνει η επέκταση, αλλά δεν θα σταματήσει τον Ιούλιο, γιατί Αυτές ε, οι διαδικασίες τώρα είναι υπό αναθεώρηση ε, και έχουμε μια δικαστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει και πρέπει να αναρωτηθούμε. Η ενίσχυση του, ε, της εκτελεστικής εξουσίας εις βάρος της νομικής ε, αυτή η ενίσχυση της αστυνομίας ε, που ξεφεύγει του δικαστικού ελέγχου είναι κάτι που μας ανησυχεί. Ε, κύριε Πρέσβη, αυτό που είπε και η συνάδελφος ισχύει. Πόσες από αυτές τις έρευνες τελικά οδήγησαν σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος, αναρωτιέμαι και εδώ στην Επιτροπή αυτό είναι το θέμα, το, θέμα μας. Συγκρίνουμε τον τρόπο που αντέδρασε η Γαλλία με αυτόν που αντέδρασε το Βέλγιο. Και στο Βέλγιο δεν υπήρξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρόλο που η απειλή της τρομοκρατίας είναι η ίδια. Ο τρόπος ε, αντίδρασης όμως δεν είναι ο ίδιος. Ε, υπάρχει επαγρύπνηση, συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας, με τον Επίτροπο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που και αυτοί αναρωτιούνται για το θέμα και εγώ πραγματικά ανησυχώ για την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μου. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει... Ο, κατάλογο έχει κλείσει και θα τον διαβάσω. Η κυρία Φαγιόν, η κυρία Ιντβέλτ, η κυρία Γκυγιόμ, η κυρία Γκόμε και η κυρία Σπινέλη. Να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για όλες τις πληροφορίες ε, που μας έδωσε ο πρέσβης ε, και πρέπει να σας πω πως ε, συμμερίζομαι πολλές από αυτές τις, πολλά από τα αισθήματα που έχουν οι Γάλλοι πολίτες λόγω των γεγονότων που λαμβάνουν χώρο. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί είναι κάτι το οποίο δημοσιεύθηκε χθε στον τύπο. Είναι από τις βελγικές εφημερίδες και από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, όπως επίσης και από κάποιους διπλωμάτες. Δηλαδή, η βελγική αστυνομία έλαβε πληροφορίες πως δύο τρομοκρατικές ομάδες έφτασαν στο Βέλιο και στη Γαλλία πριν από περίπου μια μισή εβδομάδα από τη Συρία μέσω Τουρκίας και Ελλάδος και πως χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για να εκτελέσουν επιθέσεις σε Γαλλία και Βρυξέλλες επόμενες ημέρες υποτίθεται πως έφτασαν χωρίς ε, να βγουν αυτές οι χωρίς να μαθευτεί, αλλά στα μίντια και από κάποιες πρεσβείες α, ε, ακούστηκαν κάποιες πληροφορίες ότι καλό είναι να μην μπαίνει κανείς συγκοινωνίες, να μην παγαίνει στα εμπορικά κέντρα και ζήτησε η βελγική αστυνομία από τις σχετικές υπηρεσίες να αυξήσουν το επίπεδο ε, συναγερμού στο ανώτατο. Ε, αυτό είναι μόνο κάποιες πληροφορίες στα μίδια, γιατί χτες το απόγευμα είδα πως η Βελγική Αστυνομία δήλωσε πως ακόμα ερευνά τις πληροφορίες αυτές και πως δεν θα έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη τόσο πολύ τα όσα δημοσιεύονται. Αλλά επειδή είχα πληροφορίες και από τις πρεσβείες, θα ήθελα να μου πείτε εάν εσείς ε, ακούτε τις πληροφορίες για αυτούς τους αλλοδαπούς μαχητές του ε, ISIS που φτάσανε πριν από μια εβδομάδα στο Βέλιο και στη Γαλλία. Uh, η κυρία Χόλμαγερ είναι η επόμενη μιλήτρια. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω το σεβασμό μου στη Γαλλία και τα συλληπιτήριά μου ε, για τις οικογένειες ε, που επλήγησαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις θα αναφερθώ στο ίδιο θέμα. Ε, συνεχώς μιλάμε για το αν ε, έγινε κάτι σωστά ή λάθος. Όμως, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Τι περιμένετε εσείς από την Επιτροπή μας, ε, ποια είναι η επιθυμία της Γαλλίας ε, τι θέλετε να κάνει η δική μας επιτροπή. Αλλάζω ε, την ερώτηση, την αντιστρέφω λοιπόν, γιατί καλύτερα ε, εσείς πρέπει να μας πείτε τι περιμένετε, καθώς εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι και η αστυνομία είναι στο πεδίο και πρέπει να αντιμετωπίσετε την πραγματικότητα και την τρομοκρατία. Να πω ότι, λοιπόν ότι μετά από τα τελευταία τρομοκρατικά επεισόδια οι αστυνομικοί διατρέχουν πολύ μεγαλύτερη μεγαλύτερο κίνδυνο στην ζωή τους. Ε, ε, αυτοί ε, οι άνθρωποι δεν ξέρουμε αν είναι σαλαφιστές ή δυνητικοί τρομοκράτες. Θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε λοιπόν κάτι. Σας ρωτάμε λοιπόν πώς είναι σε κατοίκον κράτηση ε, γιατί, γιατί ε, θα θέλαμε να δούμε πόσοι είναι σε θέση να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, αν ξέρετε τα ονόματά τους, ε, ποιες είναι οι στρατηγικές, υπάρχουν νέες στρατηγικές σε σχέση με αυτά τα άτομα, ε, ε, διότι υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά, αλλά είναι γνωστοί αλαφιστές. Ε, επίσης, ε, σωστά, η, η συνάδελφος ε, Φαγιών είπε ότι υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιοι τρομοκράτες που έρχονται από την Τουρκία και την Ελλάδα. Πώς πέρασαν στα ελληνικά σύνορα, τι ξέρετε, έχουμε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική σχετικά με τις οδούς που ακολουθούν οι άνθρωποι αυτοί για να εκπληρώσουν τους στόχους τους, γιατί υπάρχουν αυτοί αυτοί οι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και αυτοί που έρχονται σε εμά για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Ε, και αυτή η βάση δεδομένων που υπάρχει για τους πρόσφυγες ε, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπως. Αυτά είναι τα ζητήματα και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστούμε κυρία Ίντφελτ, έχει το ρόλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Περέσβη που ήρθατε. Νομίζω ότι ήταν σωστό και δίκαιο να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ. Ε, αντίθετα με την τόση είπε η συνάδελφος, να πω ότι ακόμα και είναι δύσκολη και δυσάρεστη η συζήτηση, τα ε, ζητήματα που συζητούμε εδώ είναι ζητήματα κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, εμείς είμαστε όλοι Ευρωπαίοι πολίτες. Οι επιθέσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο μας άγγιξαν όλους προσωπικά. Ε, όταν βλέπουμε τις εικόνες, όλος ο κόσμος κατανοεί τι συμβαίνει, το αίσθημα που επικρατεί, το συνέστημα. Ε, εκ μέρους λοιπόν της ομάδας μου θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τα θύματα και, ε, στα θύματα και στους συγγενείς τους. Να πω λοιπόν ότι μετά από κάθε επίθεση μας ζητούν να περάσουμε νόμους κατά των τρομοκρατών. Ε, δεν ξέρω πώς γίνεται ταυτόχρονα να προσέχουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εφαρμογή αυτών των νόμων, ειδικά εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Έχω λοιπόν συγκεκριμένα ερωτήματα. Ε, από την εφαρμογή με διάταγμα του κατάστασης έκτακτης ανάγκης τη 13η Νοεμβρίου του 2015 έγινε τρεις φορές παράταση, επέκταση αυτή αυτής της κατάστασης, ε, άρα ε, το καθεστώς αυτό ισχύει εδώ και 7 μήνες. Θα γίνει επιπλέον παράταση μετά τον Ιούλιο. Τι σκοπεύει να κάνει η Γαλλία. Δυστυχώς επίσης δεν είναι το πρώτο κύμα τρομοκρατίας που έχει χτυπήσει τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχει λάβει η Γαλλία ε, τα παρόμοια μέτρα στο παρελθόν σε παρόμοιες επιθέσεις. Ε, τρίτον, λέτε ότι όλα είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει ανησυχία, όμως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Συμβουλευτική Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν εκφράσει ε, μεγάλη, μεγάλες επικρίσεις. Ε, ποια είναι η κατάσταση. Επίσης, μιλήσατε για την επίσκεψη της Επιτροπής της Βενετίας. Θα ήθελα πολύ να μάθω ποια ήταν τα συμπεράσματα. Τέλος, και ίσως αυτό να είναι και ένα ερώτημα που θα έπρεπε περισσότερο να απευθύνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί λέει ότι όλα πάνε καλά, δεν μας αφορά το θέμα, είναι τελείως εθνικό. Ε, όμως, αν ε, έρθουν και άλλα κράτη-μέλη και πάρουν παρόμοια μέτρα, ας πούμε η Πολωνία, όπου ταυτόχρονα η Κομισιόν διαπιστώνει ότι υπάρχει έλλειμμα το συνταγματικό δικαστήριο δεν λειτουργεί σωστά. Τι σκοπεύει να κάνει σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν. Θα υπάρχει προηγούμενο με αυτή την κατάσταση. Και τέλος, όσον αφορά την κράτηση κατοίκων, αν κατάλαβα, αποφασίστηκαν χωρίς ε, την ε, παρέμβαση των δικαστικών αρχών ήταν ένα λευκό γράμμα που δόθηκε από τις, ε, υπηρεσίες, ε, τις μυστικές υπηρεσίες και ε, η ερώτησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατά πόσο αυτό συνάδει με το κεκτημένο το ευρωπαϊκό, το οικονομικό δίκαιο και το δικαίωμα άμυνας, το δίκαιο που έχει να κάνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αν το κατάλαβα σωστά και το τεκμήριο αθωότητας. Ε, δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί είναι υπόπτοι για τρομοκρατία ε, ή απλώς διαμαρτύνονται κατά του εργατικού δικαίου, ε, ας πούμε. ευχαριστώ. Κυρία Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μας για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ωραία, και είχα εγώ την ατυχία ναι, μια επόμενη. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που έγινε αυτή η συζήτηση. Θα τα πω στα γρήγορα και να σας πω πως είμαι από αυτούς που ήταν πολύ επικριτικοί για το θέμα του συντηγματικής διάστασης κάποιων από αυτών των στοιχείων στα οποία εσείς αναφερθήκατε σήμερα. Και είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι που δεν φτάσατε μέχρι το τέλος γιατί στα πλαίσια αυτής της ανταγματικής παράδοσης, Πιστεύω πως ε, δεν θα πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα ε, ενός ιστερικού διαλόγου του θέματος αυτού. Θα πρέπει οι συζητήσεις μας να αποφασίσουν επίσης τι γίνεται ε, επί της ουσίας. Δηλαδή, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε, να προλάβουμε και να ερευνήσουμε όπως είπατε. Οι ερωτήσεις μας είναι πολύ Συγκεκριμένε, Μιλάμε για τζαμιά τα οποία είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικοποιημένα. Όλοι έχουμε αντιμετωπίσει και δει αυτά τα βίντεο που κυκλοφορούν. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν εκεί τι πρόκειται να γίνει. Και το δεύτερο είναι, αναρωτιέμαι τι γίνεται με αυτή την κατάσταση πηγούσα ανάγκη και αν ο νόμος που ψηφίστηκε επιτρέπει να κάνουμε, για παράδειγμα, α, α, αντιπαράσταση α, τη στιγμή της ανάκρισης για να είμαστε σίγουροι για τα αποτελέσματα αυτής. Επόμενος ομιλητής. Κυρία Γκόμες, παρακαλώ. Μιλάμε για έκτακτη ανάγκη, για επίγουσα ανάγκη. Αλλά ξέρουμε πως οι απειλές στις οποίες αντιμετωπίζουμε είναι μακροπρόθεσμες. Είναι αυτή η μοναχική λύκη. Είναι χαμηλού κόστους. Είναι επιτόπου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν ήδη επιτεθεί. Για παράδειγμα, έχουμε τις ε, επιθέσεις κατά των αστυνομικών, το να μιλάμε για αλλοδαπούς μαχητές ουσιαστικά θολώνει την κατάσταση επίπεδο κοινωνικής γνώμης. Δηλαδή, μια και η απειλή αυτή είναι μακροπρόθεση, μακροπρόθεσμη και θα συμβιώσουμε μαζί έτσι για πολύ χρόνο. Κάνουμε αρκετά κατά, του, κατά της για παράδειγμα στις φυλακές, γίνονται επενδύσεις από τις κυβερνήσεις μας. Και θα ήθελα να μου πείτε και το εξής. Γιατί ανησυχείτε. ανησυχείτε για παράδειγμα το επίπεδο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τώρα, το Ορλάντο, πυροβόλα όπλα. Ξέρω πως πολλοί ενοχλούνται εδώ γιατί στηρίζουν το λόμπι των συλλεκτών όπλων. Για τους κυνηγούς για παράδειγμα κτλ. Αλλά το θέμα των πολυβόλων όπλων είναι ένα το οποίο ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ε, πολύ σημαντικό και επειδή μιλάμε για τους ασαλαφιστές, γιατί δεν κάνουμε κάτι σε, σε επίπεδο εξε, εξωτερικής πολιτικής. Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ' όλα αυτούς που διαδίδουν αυτή την εξτρεμαστική εκδοχή του Ισλάμ, όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία. Euh, euh, Είχαμε ε, αυτή τη βδομάδα μια επίσκεψη στο Κλειό και του είπαμε, οκ, αυτή τη στιγμή καταδικάζουμε τη σχέση Τουρκίας με ομάδες σαν Άρα λοιπόν, γιατί οι ευρωπαϊκές ε, ε, ε, κυβερνήσεις δεν ανησυχούν για αυτή τη διάσταση και μας είπε τότε πως ίσως θα έπρεπε. Η κυρία Σπινέλη παρακαλώ, επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Για την περιγραφή αυτή που μας κάνει της κατάστασης υπηούσας ανάγκης και των προβλημάτων που δημιουργεί. Καταλαβαίνω απόλυτα τα προβλήματα που δημιουργούνται και η χώρα μου η Ιταλία είχε μία αντίστοιχη εμπειρία της ε, δεκαετία του 70 και όπως επίσης τη δεκαετία του 80. Ε, και το τι είχαμε κάνει τότε και εμείς με το στρατιωτικό νόμο κτλ. Να σας πω πρώτα πως όταν παρατείνεται αυτή η κατάσταση επίγουσας ανάγκης, ε, τελικά δημιουργεί ένα τέρας. Γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ θεμάτων που δεν θα έπρεπε να συγχέονται. Για παράδειγμα, γίνεται μια ανάμειξη του χώρου της κοινωνικής και της πολιτικής του, του κουβίου και επίσης είναι μια κατάσταση εξαιρετική η οποία όμως διονύζεται και χρονίζει και σταδιακά αυτή η έκτατη ανάγκη περνά στο κοινό δίκαιο και αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη και στην Γερμανία και στην Ιταλία. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να μας πείτε τι σκέφτεστε γι' αυτό. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω τι πιστεύετε για την έκθεση της 9 η Ιουνίου της Ομοσπονδίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξέδωσε μια έκθεση με πολύ πολύ ανησυχητικές δηλώσεις για αυτή την ε, κατάσταση επίγουσας ανάγκης, όπου μιλάει για την κοινωνική συνοχή της χώρας και τις αρνητικές επιπτώσεις, όπως επίσης και για αυτή την ε, δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται πάνω από τους μουσουλμάνους πολίτες, όπως επίσης και βέβαια την αύξηση της λαμοσφοβίας στη Γαλλία. Μιλάμε επίσης για επιπτώσεις που δεν είναι πάντα χρήσιμες, το έχουμε πει αυτά άλλωστε, Πολύ λίγες περιπτώσεις αποκαλύψαμε κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών κατοίκου ε, που να σχετίζονται με την τρομοκρατία. Τουλάχιστον στα όσα έγινε μεταξύ Νοεμβρίου και Μαΐου μόνο 25 υποθέσεις που συγχέονται και οι 21 περιπτώσεις που γινόταν ε, απολογία του, της τρομοκρατίας. Σας καταλάβαμε κύριε μου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και ένα τελευταίο. Όταν μιλάω για αυτή τη σύγχυση μεταξύ διαφόρων θεμάτων, ζω στο Παρίσι και ανήσυχω πάρα πολύ για την ε, σύγχυση αυτή μεταξύ των κοινωνικών συγκρούσεων και της τρομοκρατίας αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπινέλη. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις κύριε Πρέσβη, θα έχετε όμως μόλις 10 λεπτά για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις, τα σχόλια, τα ερωτήματα εκ των προτέρων. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί θα είμαι πολύ ακριβή στις απαντήσεις μου όπως θα έπρεπε. Ε, μία ερώτηση που έκαναν πολλοί είναι η, ε, η διάρκεια ε, του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. με αυτό το διπλό κίνδυνο που ανέφερε και η κυρία Σπινέλη, ότι δηλαδή η εξαίρεση θα γίνει κανόνας και από την άλλη, πολλοί από εσάς Αναφέρθηκατε στην απώλεια αποτελεσματικότητας αυτού του μηχανισμού όταν θα γίνει πλέον κάτι μόνιμο. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι μια κατάσταση κατεξαίρεση, όπως είπα, ένα καθεστώς με περιορισμένη διάρκεια, όμως αυτό ταυτόχρονα πρέπει να το συμβιβάσουμε με αυτό που είπε πριν από λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός μας, ε, ότι ε, η μάχη κατά του τζιχαντισμού θα είναι θέμα μιας ολόκληρης γενιάς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η λογική του προσωρινού, της εξαίρεσης, όμως ταυτόχρονα μονίμως ε, σε πραγματικό χρόνο υπάρχει αυτή η απειλή, αυτός ο κίνδυνος ε, και υπάρχει και η κρίση από την πλευρά των αρχών που εκπροσωπώ ότι αυτή η απειλή δικαιολογεί αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί. Το δεύτερο κομμάτι της απάντησης σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει πάντοτε να υπογραμμίζουμε πως το καθεστώς έκτακτης ανάγκης είναι μια εξαίρεση και αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται το κράτος δικαίου που παραμένει ο κανόνας. Ε, απλώς υπάρχει μια προσαρμογή ανάλογα με τις καταστάσεις. Είναι πολύ ε, στόχοθετημένο ε, και να πω ότι πρόκειται για μια μόνιμη ε, προσπάθεια από τη μία να συμφιλιώσουμε τις, ε, την προστασία των ατομικών ελευθεριών και από την άλλη να, το τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να εξισορροπήσουμε αυτά τα δύο και κάθε φορά η ζυγαριά ε, γέρνει προς τη μία ή την άλλη πλευρά ανάλογα με το πώς ε, έχει η κατάσταση. Αυτή λοιπόν ε, η άσκηση, αυτή η δημόσια ευθύνη που όλοι αντιμετωπίζουμε μας αναγκάζει να θέσουμε σε ισχύ μέτρα και η Επιτροπή σας με ρώτησε κατά πόσο ε, σύμφωνα με τα νομικά ε, κείμενα ε, η ισορροπία αλλάζει κάθε φορά. Πώς δηλαδή κρίνουμε πού θα γύρει η προς την προστασία των δικαιωμάτων ή προς τα μέτρα ασφαλείας. Τρίτο στοιχείο της απάντησης. Πέρα από όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται και είναι πιθανά σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης και που πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση και την απειλή, Υπάρχει ένα παράδειγμα για να δείτε πώς ακριβώς προσαρμόζονται, πώς έγινε σε διάφορες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι κάτι σταθερό και που δεν εξελίσσεται. Για παράδειγμα, τον Νοέμβρη η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ε, ενεργοποιεί πλέον τη διοικητική έρευνα ε, για τις περιπτώσεις που έγινε αυτό στην πρώτη κατάσταση ε, έκτακτης ανάγκης. Γιατί οι περισσότερες διοικητικές έρευνες που ήταν αποτέλεσμα αποτελεσματικά, αποτελεσματικές ε, και είχαν και ένα λόγο έγιναν στην πρώτη αυτή ε, περίοδο. Ε, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ε, πρέπει να έχουμε και μακροπρόθεσμες ε, δράσεις σε βάθος που θα αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια, την ριζοσπαστικοποίηση. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που διαδίδουν όλες αυτές τις ιδέες, ε, ποιοι ε, υποκινούν αυτές τις τρομοκρατικές δράσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν να πω ότι και πολλά άλλα ε, ερωτήματα τέθηκαν, ας πούμε, από την κυρία Φαγιόν σχετικά με τον κίνδυνο άφηξης σε ευρωπαϊκό έδαφος νέων δραστών ή δυνητικών δραστών. Να επιμείνω λοιπόν ε, στη σημασία των δράσεων που από κοινού έχουμε θεσπίσει σχέση με ε, την προστασία ε, του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Σέγγεν, ε, με τον έλεγχο της εισόδου και εξόδου και πιο συγκεκριμένα είναι οι περιπτώσεις που αναφέρατε, κυρία μου, ε, πιθανές αφήξεις τρομοκρατών από την, μέσω, από την Τουρκία μέσω της Ελλάδος τα ε, διάσημα hot spot πρέπει να έχουν ε, την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν την απάτη σε επίπεδο εγγράφων και τα προγράμματα επανακατάστασης ε, που έχει ξεκινήσει βάσει της συμφωνίας που υπάρχει με την Τουρκία από τον Μάρτι να μας επιτρέπουν να κάνουμε ελέγχους ασφαλείας ήδη από την Τουρκία για να αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους που αναφέρατε. Πέρα από τον έλεγχο των συνόρων ε, που ε, έχετε εσείς αρμοδιότητα. Υπάρχει και η μάχη κατά του εμπορίου των όπλων ε, και των ναρκωτικών που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ξέρουμε ότι μετά τις επιθέσεις του Παρισιού αλλά και των Βρυξελών διαπιστώθηκε η έλλειψη χνηλασιμότητας και ελέγχου αυτών των πυροβόλων όπλων. Μετά από τις επιθέσεις στο Σαρλί η χώρα μου πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει από την Κομισιόν μια ενίσχυση της οδηγίας για τα όπλα. Το Συμβούλιο κατάφερε να έχει μια συμφωνία πριν από μερικές ημέρες και από την πλευρά των Γάλλων ε, χαιρόμαστε διότι αυτή επιτρέπει και ε, βελτίωση της περιμέτρου των απαγορευμένων όπλων Βέβαια αναφέρονται και κάποιες, χρήση, ε, κάποιες χρήσεις που είναι νόμιμες για τα πυροβόλα όπλα, ας πούμε, για τους κυνηγού ε, και τους αθλητές. Ήταν δύσκολη η διαπραγμάτευση, νομίζω ότι το ξέρει και το κοινοβούλιο σας, όμως είναι ε, απαραίτητο να βελτιώσουμε σε αυτό το επίπεδο την ιχνηλασιμότητα, τη δυνατότητα να μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κίνηση των όπλων στην Ευρώπη, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ένα κενό σε αυτό το επίπεδο. Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας επίσης είναι πολύ σημαντική, ακόμα και αν πολλές φορές ε, ε, ε αυτοί που ασκούν τις επιθέσεις δεν χρησιμοποιούν πολύ εξεζητημένα όπλα και ε, πολλές φορές ε, ε, δεν φαίνεται να υπάρχει πολύ σημαντική χρηματοδότηση απ' έξω, όμως υπάρχει χρηματοδότηση μέσω του εμπορίου όπλων, ναρκωτικών ή έργων τέχνης. Όλες αυτές οι τεχνικές πρέπει να αντιμετωπιστούν. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση και η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα ε, ένα τέτοιο σχέδιο δράσης ε, γιατί ε, έχει ήδη εξεταστεί η οδηγία για το ξέπνομα μαύρου χρήματος που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο. Άρα η συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας αυτά τα όπλα που θα μας βοηθήσουν να λάβουμε, αναλάβουμε μακροπρόθεσμη δράση, να σταματήσει αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα μας επιτρέψει να ξεριζώσουμε αυτή τη μάστιγα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτή την... Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρέσβη, για αυτή την παρουσίαση. Κυρία Ιντβελτ, πολύ σύντομα, γιατί έθεσα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας. Να σας απαντήσω και σε αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, το πόρισμα της έκθεσης της Βενετίας νομίζω δημοσιεύτηκε από την ίδια 6 Μαρτίου του 2016. collègues, nous devons passer au deuxième point de notre ordre du jour, mais on attend Madame Ferrara qui va venir dans quelques minutes, je pense. Και τώρα θα περιμένουμε για το επόμενο θέμα, γιατί η συγκήτρια θα έρθει σε λίγα λεπτά. Συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε μόνο 15 λεπτά για την έκθεση της κυρίας Φεράρα. Θα έρθει από στιγμή σε στιγμή. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτα απ' όλα, να δώσω το λόγο στον κύριο Μέλου. Κύριε Μέλου, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, για να είμαι ειλικρινής, νόημα θα είχε να δίναμε πρώτα το λόγο στην κυρία Φεράρα πρώτη, για να ακούσει και τα σχόλιά μας. Εκείνη είναι η συγγήτρια, εκείνη θα αποφασίσει ποιε είναι οι συμβαστικέ που έχουν ε, μεγαλύτερη σημασία. Ε, δεν μπορώ να κάνω σχόλια στον αέρα. Η κυρία Φεράρα είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα, οι υπόλοιποι συνάδελφοι όχι. Αυτή την πρόταση ήθελα να κάνω, αλλά αποφασίζετε εσείς κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μέλου, και εγώ την ίδια μέρη με εσάς έχω. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια και θέλω και εγώ να ε, περιμένουμε την κυρία Φεράρα, αλλά θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη και το σημείο. Το δούμε ίσως την επόμενη φορά ή σήμερα. Δεν γίνεται, διότι η κυρία Φεράρα είναι στο δρόμο. Μου είχε πει γραμματεία σε λίγα λεπτά. Euh, Η γραμματεία μου είπε να περιμένουμε ακόμη πέντε λεπτά, ιδάλλως την έκθεση της κυρίας Φεράρα, θα την δούμε, της κυρίας Λάουρα Φεράρα, θα την δούμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Η κυρία Φεράρα έφτασε. Κυρία Φεράρα, σας περιμένουμε όλοι διακαώς για να παρουσιάσετε την έκθεσή σας για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Έχετε όμως 10 λεπτά μόνο, γιατί αργήσατε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση αλλά μου είχαν πει ότι θα είναι το θέμα μου στις 10 και και όχι στις 10, με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπάβαλαν τροπολογίε. που εμπλούτησαν την έκθεση με τις συνεισφορές τους και συμμετείχαν σε όλες τις συζητήσεις για τη σύνταξη της ε, έκθεσης. Θέλω σε αυτή τη φάση να παρουσιάσω τις τροπολογίες και οφείλω να επαναλάβω μια αρχή που ήδη έχω εκφράσει και στη φάση παρουσίαση της έκθεσης και ε, όταν συζητούσαμε με τους συναδέλφους. Δεν ήθελα να πλατιάσουμε πολύ στην ε, έκθεση και στα σημεία που θα καλύψουμε. Ήθελα η διάρθρωση να είναι αυτή που είχαμε συμφωνήσει και αρχικά. Ιδάλλως, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα όπως και με το ψήφισμα της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Θα είναι λίγο τόσο, θα είναι τόσο ευρεία που θα είναι σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, θα τα περιλαμβάνει όλα. Πολλές τροπολογίες υποβλήθηκαν και εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου που θέλαμε να παρέμβουμε της αρχικής μας πρόθεσης, ήταν τροπολογίες σημαντικές, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη και Σίγουρα κάποια πράγματα χρειάστηκε να προστεθούν όπως η παραποίηση φαρμακευτικών, και, τροφή, φαρμακευτικών προϊόντων και τροφίμων, οι δημόσιες προμήθειες. Είναι συγκεκριμένα σημεία στα οποία χρειάστηκε να παρέμβουμε και όντως εμπλούτησαν την αρχική έκθεση. Όμως, όπως έλεγα και προηγουμένως, για να, για να γίνει ε, πιο συγκεκριμένη η έκθεση. Θα φροντίσουμε να υποβάλουμε και συμβιβαστικέ λύσει, συζητώντα με του κοιόδη συναδέλφου, ώστε να ομαδοποιήσουμε όσο γίνεται τι τροπολογίε και να παραμείνει η δομή με συγκεκριμένου στόχου. Προτάθηκαν πάρα πολλέ τροπολογίε, ενδιαφέρουσε, για του πληροφοριοδότε, για του συνεργάτε της δικαιοσύνη, και τη δικαστική του προστασία, για την εισαγγελία την θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, αλλά κάποιες φορές ε, δυσανάλογα σε σχέση με άλλα θέματα που καλύπτει η έκθεση. Οπότε, για λόγους εξισορρόπησης μεταξύ των διαφορετικών θεμάτων που ε, καλύπτει η έκθεση και για να έχουμε συγκεκριμένη δομή με συγκεκριμένους στόχους, θα κοιτάξουμε να τα ομαδοποιήσουμε για να είναι και βανάγνωστη η έκθεση. οι τροπολογίες για τις κλιματικές οργανώσεις τύπου μαφίας, για την διαφθορά, είναι τροπολογίες οι οποίες θα κοιτάξουμε να συμπεριληφθούν, αλλά θα σταματήσω εδώ για να ακούσω και τους συναδέλφους και να σεβαστώ και το χρόνο που μου δώσατε τα δύο λεπτά. Ευχαριστούμε και τώρα κύριο Μέλου, έχετε το λόγο για δεύτερη φορά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο Φεράρα για τη δουλειά της και τις προσπάθειές της. Εργάστηκε σκληρά για μια έκθεση που είναι σημαντική λόγω του θέματός της και που ενδιαφέρει ολόκληρη την Ευρώπη. Με όλους τους κοιόδης εξηγητές, αλλά εγώ θα μιλήσω προσωπικώς. Ε, νομίζω ότι δείξαμε μεγάλη αφοσίωση και υποβάλαμε ένα σύνολο τροπολογιών που θα ήθελα να τις αντιληφθεί η συνάδελφος ως θετική συνεισφορά στο τελικό αποτέλεσμα και να τις αξιοποιήσει σε διάφορους τομείς της, ε, δημο, της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ξέρουμε ότι είναι τομείς που είναι ευάλωτοι στην ε, ε, διαφθορά, τις δημοτικές αρχές, την ε, εθνική διάσταση της διαφθοράς, αλλά πολλές φορές αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειών, της, την διαφθορά στη, στον αθλητισμό και στις αθλητικές εκδηλώσεις. Ξέρουμε ότι κάποιες φορές μας εκπλήσουν αυτά που ακούμε στα νέα. Το τι γίνεται με τα λόμπι, τις ομάδες άσκησης πίεσης. Ε, σίγουρα είναι νόμιμη η δράση του, αλλά πρέπει να διαθετηθεί για να αποφύγουμε καταστάσει που να μην είναι σαφείς. Το θέμα των νέων τεχνολογιών που επιβάλλουν όποιο κάνει ανακρίσει για εγκλήματα να έχει τα απαραίτητα οικονομικά, τεχνολογικά και υλικά μέσα για να μπορεί να κάνει τις ανακρίσεις και τις έρευνες που χρειάζεται. Πολλές αστυνομικές αρχές δυσκολεύονται να εντοπίσουν την μεγάλη κλίμακα της οικονομικής διαφθοράς που έχει διασυνοριακό χαρακτήρα και δεν μπορεί να καλύψει με το προσωπικό που διαθέτει. Επίσης, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, διότι δεν έχουν όλα τα, κόμματα, τους ίδιους, όλα τα κράτη του ίδιου κανόνε για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Θα πρέπει αυτό να το δει το Κοινοβούλιο και μερικά λόγια για τους πρόσφυγες. Ε, εκμετάλλευση του ανθρώπου. Και κάποιοι εκμεταλλεύονται το ίδιο το φαινόμενο. διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα οικονομικά και είναι τα οικονομικοί λόγοι. Πρέπει και αυτά να καταπολεμηθούν. Και επίσης ο χώρος ε, έρευνας και ανακρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τι είναι εξωτερική έρευνα και το τι μπορεί να συμβαίνει εξωτερικός. Μπορεί να έχουμε πολλούς ε, θυγόμενους από τέτοιες έρευνες και ενδιαφερόμενους που για αυτά τα θέματα θα πρέπει να αναπτύξουμε μια ε, προσέγγιση σφαιρική. Η δική μας πολιτική ομάδα λοιπόν θα συνεισφέρει στην ε, εκπόνηση της έκθεσης αυτής με όσο πιο θετικό τρόπο γίνεται και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για όλο το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Μέλου. Ως ε, σκιώδης εισηγήτρια θα μιλήσω βουλγαρικά και θα πω λίγα λόγια και εγώ για αυτό το θέμα. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω κυρία Φεράρα για αυτή την τόσο καλή γνωμοδότηση που ήταν πραγματικά... Ε, πολύ ενδιαφέρουσα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι πρότειναν τροποποιήσεις και τροπολογίες. Θα μπορούσα να κάνω μία σύγκριση γιατί κατά την ε, προηγούμενη θητεία ασχολήθηκα με την έκθεση για κουλίνο και η έκθεση αυτή είχε ως σκοπό να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για την διαφθορά, το ξέβλημα χρήματος και το οργανωμένο έγκλημα, κάποια μέτρα κατά πολέμησης αυτών. Σύμφωνο με την κυρία Φεράρα, θέλουμε μια πιο στοχευμένη έκθεση και θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με κάποιες διαστάσεις του θέματος. Αυτή τη στιγμή καλύψουμε ένα ολόκληρο φάσμα και στη δουλειά που κάναμε ε, και στην προηγούμενη έκθεση καλύψαμε όλα αυτά τα θέματα και όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρουσίασε και δεν κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις. Θα ήθελα όμως να πω πως η έκθεση Φεράρα ήταν πολύ πιο συγκεκριμένη και θεωρούμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τη διαβάσει και να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις βασιζόμενες σε αυτήν. Και επειδή εδώ εκπροσωπώ και κάποιους άλλους συναδέλφους από τους σοσιαλιστές, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις τροπολογίες μας, όχι βέβαια κάθε μία από τις τροπολογίες, γιατί χρειάζεται να εξοικονομήσουμε χρόνο, αλλά Θα ήθελα καταρχήν να σας κάνω κάποιες προτάσεις για τους διαφορετικούς μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχω το, τη CVM εδώ κατά νου καταρχήν και θα έπρεπε ε, να έχουμε και το ε, scoreboard για την δικαιοσύνη και όλα αυτά ε, να τα εφαρμόσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη με πιο διευρυμένο τρόπο. Ξέρετε πως η μία έκθεση που λάβαμε και την οποία συνέταξε η Κομισιόν ε, δίνει πληροφορίες για το τι κάνουν τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της διαφοράς και αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα σε όλα τα κράτη-μέλη με το θέμα αυτό. Δεύτερον, έχουμε κάποιες τροπολογίες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς στις, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κάποιες τροπολογίες οι οποίες σχετίζονται με την ανάγκη εναρμόνισης των διαφόρων νομικών διατάξεων που ισχύουν στο ποινικό δίκαιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την εισηγήτρια και πιστεύω πως ε, θα πετύχουμε τους απαραίτητους συμβιβασμούς και θεωρώ πως οι δικές μας τρολογίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενταχθούν στο κείμενο. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, θα δώσω το λόγο στην κυρία ε, Γκρισμπέκ από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε χρόνο, να ευχαριστήσω τη Λάουρα για την πολύ καλή δουλειά, τη συνεργασία, τη συναντήσεις, την ανταλλαγή απόψεων. Το είπα ε, την τελευταία φορά που συζητήσαμε αυτό το θέμα ότι είχε μια πολύ καλή ιδέα και μπόρεσε να ε, οργανώσει ανταλλαγή απόψεων με ε, επαγγελματίες για το θέμα το εισαγγελικό. Σύμφωνα λοιπόν <clears throat> ε, με αυτά που έχουν υποθεί δύο υπάρχουν τέσσερα σημεία στα οποία επιμένουμε. Βλέπουμε ότι είναι διεθνικό το, η διεθνική δράση των ε, εγκληματικών οργανώσεων και γιατί δρούν σε πολλές χώρες. Για να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει με επίγον τρόπο να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία που θα μας αποτελέσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είμαστε αποδοτικοί αποτελεσματικοί. Χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν που θα έχει τους απαραίτητους πόρους και μία εντολή, μία αποστολή που δεν θα περιορίζεται στα οικονομικά προβλήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, γιατί η αποτελεσματικότητα της μάχης κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος δυστυχώς πάσχει από έλλειψη συνεργειών ε, όσον αφορά στις δράσεις που αναλαμβάνονται για το συγκεκριμένο σκοπό. Χρειάζεται λοιπόν μια συστηματική δυνατότητα χρήσης ε, των βάσεων δεδομένων ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτόματα συστηματικά να μπορούν η Ευρωπολή, η Eurojust, η Eurojust και όλοι αυτοί οι οργανισμοί να συνεργάζονται. Επίσης είναι πολύ σημαντικό δεδομένου του οικονομικού βάρους ε, του ξεπλήματος χρήματος και της παραποίησης να ε, επανέλθουμε στο θέμα του οργανωμένου εγκλήματος ε, και να επιμείνουμε σε αυτό για να μπορέσουμε να ε, βελτιώσουμε κάθε μορφή μάχης κατά της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Για την κατάσχεση αγαθών να πω ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια προσπάθεια υπό την αιγίδα της Λάουρα Φεράρα να γίνει μία αναθεώρηση της οδηγίας μέσω, του, μέσω της οποίας θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να διώκουμε άτομα τα οποία μεταφέρουν την κυριότητα των ε, πάγιων στοιχείων τους για να μπορέσουν ε, να αποφύγουν την κατάσχεση. Τα δίνουν δηλαδή σε μέλη της οικογένειάς τους κτλ. Να έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτές οι μεταβιβάσεις να μην επιτρέπονται. Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν αποκτηθεί με εγκληματικό τρόπο. Και επειδή πάντοτε σε αυτήν την Κομισιόν πρέπει να βιαζόμαστε, ε, να πω ότι θα τελειώσω, αλλά να πω ε, ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις βάσει αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ κυρία Γκρίσπεκ και τώρα Κύριος Ντεγιόγκ, ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα είμαι πολύ σύντομο γιατί πρέπει να τρέξω σε άλλη επιτροπή σε λίγα λεπτά. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις συζητήσεις που είχαμε, τις πολλές ε, άτυπες ε, συνεννοήσεις, συνεδρίασεις συντονιστών. Συμφωνώ με τη γενική προσέγγιση κατά πολύ η έκθεση να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένη γίνεται και πιο σαφή για να αποφύγουμε καταστάσεις όπου η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα καταλήξουν να μας πούν τι ωραία έκθεση του Κοινοβουλίου, αλλά θα πάρουμε μόνο ένα-δυο στοιχεία και τα υπόλοιπα θα τα πετάξουμε. Τα ξεχνάμε. Ε, πρέπει να έχουμε ένα πλήρες σύστημα συστάσεων στο ψηφισμά μας, που θέλουμε η Επιτροπή και το Συμβούλιο να τα λάβουν σοβαρά υπόψη ενός αντικείμενο σχεδιαζόμενης δράσης για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε τη δική μου ομάδα, ο τέλο πάντων γενικώ τι τροπολογίε, θα τονίσω ένα θέμα, την τροπολογία 34, γιατί είναι αρκετά μοναδική στο είδος της, είναι μια υπενθύμηση των γενικών αρχών που ήδη έχουμε εγκρίνει ω Κοινοβούλιο για το ποινικό δίκαιο, το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και την ευρωπαϊκή του διάσταση και πρέπει να θυμόμαστε εδώ ότι κάποια κριτήρια όταν προβλέπουμε νέα νομοθεσία στο ποινικό δίκαιο, ισχύουν υποχρεωτικά. Στην έκθεση αυτή έχουμε προσέξει τη διάσταση αυτή. Και κατά δεύτερον, να εξηγήσω ότι μέρος της των τροπολογιών που βλέπετε το όνομά μου, μαζί με συναδέλφους βουλευτές από άλλες πολιτικές ομάδες, αυτά αντικατοπτρίζουν τη θέση της ε, διατομιακής ομάδας για τη διαφάνεια κατά της διαφθοράς, την λεύκανση ε, χρήματος και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε κοινέ απόψεις που ούτως ή άλλως έχουν διαμορφωθεί μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων στην διακομματική ομάδα εργασίας μας και με σκοπό να διευκολύνουμε την δουλειά της ε, εισηγήτριας και την εξέβριση συμβαστικών τοπολογιών. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόν, ο κύριος Τερικάμπρας, αν σωστά προφέρω το όνομά σα από τους πράσινου σωστά. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λάβει το λόγο εκ μέρου τη Εύα Ζολή, η οποία δυστυχώς δεν είναι σε θέση να παραστεί σήμερα. Θα είμαι πολύ σύντομο και εγώ πρέπει να φύγω, θα τα πω λοιπόν στα γρήγορα. Εγώ πάντα επιμένω στα εξή σημεία. Η τροπολογία 155, για παράδειγμα, τονίζει πως ο αριθμός των περιβαλλοντικών εγκλημάτων αυξάνεται και πως θα πρέπει να απευθυνθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνοντας πλήρως υπόψη ε, της, ε, τη σύνδεση που έχει με εγκληματικές οργανώσεις τύπου μαφίες. Οι τροπολογίες 94 με 98 ε, υπογραμμίζουν το βασικό ρόλο που έχει να παίξει το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την κατάταξη της διαφθοράς στην Ευρώπη. Ε, θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε να έχουμε έναν εξάρτητο και ισχυρό γραφείο Ευρωπαϊκή εισαγγελία με ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Επίσης, κάποιες από τι τροπολογίε μας έχουν σκοπό να ασκήσουν πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταθέσει προτάσει για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Γιατί αυτοί ακριβώ οι πληροφοριοδότες παίζουν μεγάλο ρόλο, που αποκαλύπτουν μυστικά, παίζουν μεγάλο ρόλο στη μάχη κατά της διαφθοράς. Ξέρετε τι έγινε με τα LuxLeaks και τα Panama Papers. Όλα αυτά ε, αποδεικνύουν πως πρέπει να δράσουμε στο χώρο αυτό. Και τέλος, η Επιτροπολογία 193 λέει στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πως θα πρέπει να παρακολουθήσει τις, κατευθυ... συστάσεις που είχαμε στο ψήφισμά μας, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ένα ψήφισμα το οποίο δεν θα έχει ισχύ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δράσεις μας στον χώρο αυτό, στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να δώσουμε σάρκα και ωστά στις συστάσεις μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Φεράρα για τη συνεργασία της εδώ γιατί είναι πολύ σαφής, σύντομη, στοχευμένη, περιεκτική και θα είναι πολύ σημαντικό να, είναι, ε, να έχει αυτή τη μορφή αν θέλουμε να ακουστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ο κατάλογος έχει κλείσει, συνάδελφε. Δύο μου ζητούν ακόμη το λόγο. Θα, θα δώσω το λόγο στην κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Φεράρα που αξιοποίησε τα πορίσματα της Επιτροπής ΚΡΙΜ και εκπώνησε το έγγραφο αυτό στο οποίο προσπάθησα και εγώ να συνεισφέρω με προτάσεις για τροπολογίες. Προφανώς το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος για το οποίο σήμερα δεν έχουμε ούτως ή άλλως ένα κοινό ορισμό και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί ένα σημείο θετηρία το οποίο πρέπει να το δούμε με προσοχή διότι όταν θέλουμε να εμβαθύνουμε στο θέμα προφανώς υπάρχουν αποκλήσεις και στην Επιτροπή μας αλλά το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και το οποίο διαρκώς εξελίσσεται και έχει λάβει χαρακτηριστικά διασυνοριακά. Γι' αυτό δυστυχώ μπορεί να δυσδύσει σε διαφορετικού τομείς και σε διαφορετικές ε, δράσει. Ε, σε διαφορετικούς τομείς δράσεις. Όπως είπε και η πρόεδρο μας Γιώτοβα σήμερα, πρέπει να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε σε μερικές πτυχές στο εγγραφό μας. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη την περιπλοκότητα αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό ε, πιστεύω σημαντικό είναι να ε, θίξουμε τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τις παρεμβολές του οργανωμένου εγκλήματος στην ε, νόμιμη οικονομία, την ένομη οικονομική δράση των κρατών μελών. Εκεί χρειάζονται περισσότερο παρεμβάσει. Ξέρουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα δυσδύει στην πραγματική οικονομία μέσω τη διαφθορά, τη ανακύκλωση, παρεμβαίνοντα σε διάφορε δραστηριότητε αναλυτικού τύπου. Χθε μόλι συζητούσα με μία συνάδελφο που μου έλεγε ότι υπάρχει δίσδυση του οργανωμένου εγκλήματο ακόμη και στον τομέα τη αλληλεία. Κάτι που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ. Είναι όμω ένα τομέα παραγωγή σημαντικό που παρόλα αυτά δυστυχώ πλήττεται από το οργανωμένο έγκλημα. Εδώ λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε ακριβώ σε αυτή την πτυχή. Ε, Εδώ λοιπόν είναι σημαντική αυτή η πτυχή και πραγματικά και εγώ συμμερίζομαι την ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται, δίνεται λόγω χάρη στην προστασία των μαρτύρων στη δικαιοσύνη. Στην Ιταλία ε, δυστυχώ και αλίμονο έχουμε γνωρίσει το φαινόμενο αυτού του οργανωμένου εγκλήματο με διαφορετικού τρόπου. Ξέρουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι και αυτή η διάσταση. Και μία τελευταία παρατηρήση, γιατί ξέρετε πρέπει να είμαι συνοπτικότατη, είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Γιατί υπάρχουν διασυνοριακά το οργανωμένο έγκλημα έχει γίνει διασυνοριακό φαινόμενο, άρα είναι θεμελιώδη και να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε ε, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο λογιστικό και οικονομικό τομέα, όπω και προηγουμένω. Είναι σημεία ισχυρά αυτά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με δραστικό τρόπο το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ευχαριστώ κυρία Κινίτσι. Η κυρία Σλέιν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια και όλου του κοιότητε εισηγητέ για αυτή την τόσο σημαντική του δουλειά Προσπάθησα να συνεισφέρω και εγώ, υποβάλλοντας κάποιες τροπολογίες που ξέρω ότι προσπαθώ τουλάχιστον να δώσουν έμφαση στα σημεία που είναι προσφυλή και στην συνάδελφο Φεράρα. Πρώτα απ' όλα, ζητώντα να υπάρξει νομοθετική πράξη η οποία να θεσπίσει κοινού κανόνες για την προστασία των πληροφοριοδοτών, whistleblowers, η οποία είναι απαραίτητη πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ελάχιστα, εξελαχίστον τουλάχιστον αναγνωρισμό και το ίδιο ισχύει και για του μάρτυρε στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια. Επίσης, οι κοινέ δηλώσεις για την έγκριση της οδηγίας ε, δημεύσεων και κατασχέσεων πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει αυτό που έχει υποσχεθεί. Ε, δηλαδή μια νομοθετική πρόταση που να αναγνωρίζει να επιτρέπεται την αμοιβαία αναγνώριση των ε, εντολών κατάσχεση και για την προστασία των κληρονομικών δικαιωμάτων και γιατί όπως πάντοτε, όπως προέβλεπαν οι δηλώσεις που έχουν προσαρτηθεί στην οδηγία για να μπορεί να δεσμευτεί και το κέρδος, ε, τα ωφέλη που μπορεί να έχουν να κάνουν με τα περιουσιακά στοιχεία που ε, δεσμεύονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το οργανωμένο έγκλημα και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την εμπειρία μας στην Ιταλία. Επίσης, το match fixing, ε, το στήσιμο ποδοσφαιρικών παιχνιδιών. Βρισκόμαστε σε περίοδο γιούρο. Πρέπει λοιπόν να ε, αντιμετωπίσουμε τα παράνομα στοιχήματα και τα στημένα παιχνίδια, τους στημένους αγώνες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που διαρκώς αντιμετωπίζουμε και προσκαλούμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σλέιν και τώρα μια μικρή εξαίρεση. Κύριε Ράντεφ, τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει ένα συγκεκριμένο κράτος. Υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση. Και γι' αυτό επιμένουμε για άλλη μια φορά ε, στην ύπαρξη μιας ευρωπαϊκής ε, στρατηγικής για τη μάχη κατά της διαφθοράς. Η μάχη κατά της διαφθοράς ε, αυτή τη φορά θα πάρει την προσοχή, θα λάβει την προσοχή που της αξίζει. Θα συνεργαστούν καλύτερα τα κράτη-μέλη μεταξύ τους και θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Έχω προτείνει μία τροπολογία βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να παρακολουθεί αυτή τη μάχη κατά της διαφθοράς σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτός ο μηχανισμός παρακολούθησης ε, μπορεί να είναι όμοιος με το μηχανισμό συνεργασίας και παρακολούθησης που υπάρχει μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά Τέλος, φαντάζομαι ότι θα υποστηρίξετε την τροπολογία μου που έχει να κάνει με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ράντεφ. Ε, να σας πω ότι θα ψηφιστεί στις 11 και 12 Ιουλίου μάλλον η έκθεση αυτή, στη συνεδρίαση δηλαδή εκείνη, είναι τελευταία συνεδρίαση πριν τι τερινέ διακοπέ και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, εφαρμογή του συστήματο των κέντρων πρώτη υποδοχή hotspot στην Ιταλία. Θα ακούσουμε τον κύριο Ονίντι. Είναι εδώ. Κύριε Ονίντι, θέλετε να έρθετε στο Προεδρείο. Όχι. Έρχεστε. Τέσσερα άτομα. Συνάδελφοι, η προσέγγιση των ε, ε, hot spot ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση. Τα κέντρα πρώτη υποδοχή που έχουν να διευκολύνουν τη διαχείριση από τα κράτη-μέλη του μεγάλου αριθμού μεταναστών που φτάνουν στα σύνορά μα στη Μεσόγειο. Στα κέντρα από τι υποδοχή, τα κράτη-μέλη και οι υπαλληλοί του, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών φορέων, σκοπό έχουν να εντοπίσουν γρήγορα, να καταγράψουν και να επεξεργαστούν τι αιτήσει ατόμων που, που χρήζουν διεθνού προστασία. Τα hotspot λοιπόν ε, είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με το πρόγραμμα επαναγκατάστασης και την ε, πραγματική επιστροφή, την ε, ουσιαστική επιστροφή, αυτό που δεν έχουν δικαίωμα στο άσυλο σε άλλη μορφή επικουρικής προστασίας. Ενώ είχαμε συζητήσει τα θέματα αυτά για τη λειτουργία των hotspot στην Ελλάδα την ε, περασμένη Δευτέρα ε, επαφορμή της ε, επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ εκεί, σήμερα θα επικεντρωθούμε στην κατάσταση στην Ιταλία που έχει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων που φτάνουν στην Ιταλία τις τελευταίες εβδομάδες. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον αναπληρωτή διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης HOME, τον κύριο Νίδη, ο οποίος πρόσφατα επισκέφθηκε τα κέντρα πρώτης υποδοχής στην Ιταλία για να μας παρουσιάσει το πώς έχουν τα πράγματα. Με μεγάλη χαρά σας υποδέχομαι στην Επιτροπή Λίμπε για πρώτη φορά από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας. Μετά από την παρέμβασή σας θα έχουμε και τις παρεμβάσεις από την υπατερμοστία του ΟΗΕ και τον εκπρόσωπό της, οπότε οι συνάδελφοι θα έχουν και την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις. Κύριε Ονίδη, δεν έχουμε πολύ χρόνο συνήθως στην Επιτροπή μας, γι' αυτό λοιπόν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την εισαγωγή. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ σε αυτή τη διαδικασία της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σας ενημερώσω για την κατάσταση των hot spots στην Ιταλία και γενικά για την κατάσταση των ε, μεταναστών ε, στην Ιταλία αλλά και τη δυναμική στο κεντρικό διάδρομο της Μεσογείου όπως ονομάζεται ο οποίος γίνεται όλο και πιο σημαντικός ειδικά μετά τη συμφωνία με την Τουρκία. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως από αυτή την οδό. Η κατάσταση σήμερα λίγο πολύ ε, έχει ως εξής. 55.000 ε, μετανάστες έχουν ε, αποβιβαστεί στην Ιταλία. Την περασμένη εβδομάδα πάνω από 6.000 διασώθηκαν στη θάλασσα και αποβιβάστηκαν στην Ιταλία. Τα ίδια τα νούμερα δεν διαφέρουν από την τάση που είχαμε συνολικά και πέρυσι. Η Ιταλία βέβαια αντιμετωπίζει την κατάσταση βάσει της εμπειρίας που έχει αποκτήσει με την πάροδο των ετών. Δεν υπήρξε αλλαγή των οδών. Ε, είναι ένα στοιχείο που συζητήθηκε σε αυτή την Επιτροπή. Δεν βλέπουμε αλλαγή των οδών που ακολουθούν οι άνθρωποι που έρχονται από την Συρία, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, αυτοί που ερχόντουσαν παραδοσιακά από αυτή την οδό, την κεντρική οδό της Μεσογείου, αυτοί συνεχίζουν να έρχονται και τώρα Νιγηριανοί ε, και άνθρωποι από την Ερυθρέα, την Αιθιοπία, τη Σομαλία, το Σουδάν κτλ. Εδώ επίσης ε, να πω ότι το 87% των ανθρώπων που ε, επιβιβάζονται σε βάρκες ε, είναι από την, το κάνουν αυτό στη Λιβύη και το υπόλοιπο ποσοστό στην Αιγυπτό. Οι άνθρωποι λοιπόν που έρχονται από την Αίγυπτο μας ε, έκαναν να προσπαθήσουμε μαζί με τις Αιγυπτιακές αρχές να λάβουμε κάποια επιπλέον μέτρα και να κατανοήσουμε γιατί αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν δύο βασικές τάσεις ε, που έχουν να κάνουν με την κατάσταση που είχαμε πέρυσι και τη σύγκριση με αυτή την κατάσταση. Έχουμε κάποια σημαντική έξαρση, ειδικά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου ε, Ε, είδαμε ε, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που μέσα σε μία μέρα αποβιβάστηκαν ε, κάτι που είναι μεγάλη πρόκληση για τις αρχές καθώς θα πρέπει να δώσουν μία στέγη σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάτι άλλο που εσείς πολύ συχνά θέτετε ως ζήτημα είναι ο μεγάλος αριθμός απολειών ζωής. Ε, έχουμε πολύ συχνά, δυστυχ... έχουμε δυστυχώς μία μεγάλη αύξηση κατά 30% στους ε, θανάτους σε σχέση με πέρυσι και ξέρουμε ότι στα τέλη του έτους ο αριθμός ε, θα αυξηθεί, θα είναι πολύ αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες ε, ως προς τις ε, διάφορες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται περισσότερο υποστήριξη. Δεν αμφισβητούμε βέβαια αυτή τη στιγμή την ε, αποτελεσματικότητα των εφιστάμενων επιχειρήσεων, όμως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι διακινητές χρησιμοποιούν χαμηλότερης ε, ποιότητας μέσα ε, πλεύσης ε, και βάζουν σε αυτά περισσότερο κόσμο. Έχουμε φουσκωτά που χρησιμοποιούνται για να φέρουν πάνω από 100 άτομα από τη Λιβύη ένα νέο φαινόμενο και όσοι άνθρωποι έρχονται από την Αίγυπτο επιβιβάζονται σε αλλιευτικά ε, σκάφη που ε, τα φέρουν πάνω από 300 άτομα. Τεράστια λοιπόν πρόκληση και για την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Ε, έχουμε τέσσερα hot spot στην Ιταλία, τα οποία λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά εδώ και καιρό ε, Λαμπετούζα, Τραπάνη, Τάραντας μεταξύ αυτών και επιβεβαιώθηκε πρόσφατα ότι θα ανοίξουν άλλα δύο και θα λειτουργούν από τον Ιούλιο. Κάτι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε ότι αυξάνονται οι αριθμοί και οι καιρικέ συνθήκες βελτιώνονται, άρα θα υπάρξει και άλλη αύξηση. Θα στο Μήνο και στη Μεσίνα, θα είναι, ε, στη Μεσίνα θα είναι αυτά τα hot spots που θα δημιουργηθούν. Επίσης, ως προς την... Ε, ε <coughs> τις Ιταλικές αρχές να πω ότι θέλουν να έχουν και, τέσσερις και τέσσερα κινητά hot spot για να μπορούν να πηγαίνουν από το ένα μέρος της Ιταλίας στο άλλο και να αυξήσουν την ε, αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ε, ε, αποβίβασης. Αυτές οι κινητές μονάδες, ας πούμε, πολύ γρήγορα θα επισημοποιηθούν, θα γίνουν πραγματικά hot spot, γιατί χρειάζεται αυτή η δυνατότητα. Τα τέσσερα κινητά hot spot θα είναι στην Αγκούστα, Παλέρμο, Ρέτζιο και στον Κρότονα. Συνολικά θα αυξηθεί από τα 1.600 άτομα στα 3.000 ή λίγο παραπάνω άτομα η ικανότητα φιλοξενίας αυτών των hot spot. Επίσης, πάνω από το μισό των μεταναστών φαίνεται ότι αποβιβάζονται εκτός των hot spot. Ξέρετε ότι αυτό ε, το μήνυμα ε, το έχετε κι εσείς ε, απευθύνει προς εμάς πάρα πολλές φορές. Χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη ε, αύξηση των ικανοτήτων γιατί ε, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης στα hot spot. Επίσης υπάρχουν αυτά τα πλευστά hot spot, πλωτά hot spots, ε, είναι μια νέα καινοτόμως ιδέα. Θέλουμε να γίνουν όλα στη θάλασσα, σε ένα σκάφος το είπατε ορμοστία για τους πρόσφυγες και οι δικοί μας οργανισμοί έχουν θέσει διάφορα ερωτήματα. Τι ακριβώς είναι αυτό. Ε, εδώ ε, πραγματικά ε, μάλλον θα υποστηρίξουμε τις Ιταλικές αρχές να τα χρησιμοποιήσουν γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε άλλο ένα ναυτικό εργαλείο ε, ένα σκάφος για 2.000 με 2.500 άτομα ε, που θα μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ε, έρευνας και διάσωσης και τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών στα κανονικά hot spot, έτσι ώστε να έχουμε 100% αποβιβάσεις σε hot spot και να μπορούμε άμεσα να δίνουμε ιατρική φροντίδα και σε και σωματική και ψυχική, και για τη σωματική και για την ψυχική υγεία των μεταναστών, ε, έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και φροντίδα των μεταναστών όταν φτάνουν στα hot spot. Γενικά οι συνθήκες στα hot spot είναι πολύ καλά καλές. Έχουμε όλες τις ε, ομάδες, των ε, Διεθνή Οργανισμών Μετανάστευσης, την Υπατερμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες που δρούν στα hot spot. Στείλαμε επιστολή στις Ιταλικές αρχές πριν από 10 μέρες ε, σχετικά με πιθανές βελτιώσεις στον υποδομή, στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι μετανάστες, που θα πρέπει να γίνουν και οι Ιταλικές αρχές τις λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Επίσης, ε, έχουμε και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης ε, που θεσπίσαμε μαζί με τις ε, Ιταλικές αρχές. Βέβαια, οι Ιταλοί από την πλευρά τους δεν θέλουν να μιλάνε για έκτακτη ανάγκη, γιατί για αυτούς η κατάσταση είναι κάτι συνηθισμένο. Όμως, με τον ε, Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την ΥΠΑΤΗ αρμοστία το ΕΕ για τους πρόσφυγες, ε, θέλαμε να δείξουμε στις Ιταλικές Αρχές ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ε, τη, ε, την μια κατάσταση κατά την οποία οι εξάσεις που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες ε, θα γίνει ο κανόνας, να μπορούμε δηλαδή να κινητοποιηθούμε γρήγορα. Ε, πολλά είναι τα ερωτήματα που απομένουν για την κατάσταση στην Ιταλία. Εχθές είχατε νομίζω με την Επιτροπή μια πολύ καλή συζήτηση σχε... βάσει της έκθεσης που εκδόθηκε χθες η Ιταλία αναλαμβάνει πολύ σοβαρά ε, τις ευθύνες της και υπάρχει ανάγκη και εμείς από την πλευρά μας να το κάνουμε και να βοηθήσουμε λίγο τους Ιταλούς. Αυτό σημαίνει ότι ο ε, μηχανισμός επανεγκατάστασης πρέπει να ε, είναι πιο αποτελεσματικός, να μην είναι μόνο υποσχέσεις. Χρειάζονται Βέβαια, ε, όλες αυτές οι διαδικασίες ε, που απαιτούνται για τους ετούντες άσυλο, ε, για τη σωστή τους αντιμετώπιση στην Ιταλία, έχουμε συνεργασία συνεργαστεί με τις ε, άλλες χώρες μέλη έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή, ε, να πάρουν τους ανθρώπους αυτούς ε, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι αυτοί μένουν πολλές φορές, πολλούς μήνες κάπου κοντά σε ένα hot spot με την υπόσχεση ότι θα φύγουν. Οι Ιταλικές αρχές έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Έχουν καταγράψει υποψήφιους. Έχουμε ας πούμε 4.000 πολίτες της Ερυθρέας που θα μπορούσαν πολύ σύντομα με πολύ μικρή ειδοποίηση να ε, πανεγκατασταθούν σε άλλες χώρες. Υπάρχουν κάποιες εκατοντάδες ε, που ε, θα μπορούσαν να προσταθούν σε αυτούς, αλλά το, ο ρυθμός είναι πολύ αργός. Μόνο 25 έφυγαν τις τελευταίες εβδομάδες. Πρέπει να γίνει λοιπόν προτεραιότητα το θέμα. Δεύτερη προτεραιότητα. Η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Δυστυχώς έχουμε δει αύξηση. Έχουμε ένα ποσοστό περίπου 12% ε, που αποτελεί ασυνόδευτους ανηλίκους. Είναι ανήλικοι, ένας δύσκολος πληθυσμός, ε, ε, δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε εύκολα. Οι Ιταλικές αρχές κάνουν πολλές προσπάθειες να φροντίσουν αυτούς τους ανθρώπους, να τους βοηθήσουν όμως εδώ χρειάζεται κινητοποίηση. Χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Χρειαζόμαστε πιλωτικά προγράμματα επανεγκατάστασης και για αυτούς τους ανθρώπους ε, ε, για να δείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε ε, καλές συνθήκες και την σωστή παρακολούθηση, το follow-up στην χώρα που θα πάνε. Αλλά χρειαζόμαστε και άλλα προγράμματα υποστήριξης. Ένα ε, συγκεκριμένα που θα έχουμε μαζί με τη UNICEF. Κάτι άλλο ε, πολύ σημαντικό ε, που έχει να κάνει με την Ιταλία είναι ότι πρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός των επιστροφών. Υπάρχουν κάποια επιτυχημένα προγράμματα που πρέπει να ξεκινήσουμε τη βοήθεια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για να μπορέσουμε και να δώσουμε μια όθηση σε τα εθελοντικά προγράμματα που ήδη ε, λειτουργούν, αλλά ε, και να αποφύγουμε τις κρατήσεις των ανθρώπων αυτών καθώς περιμένουν την μετεγκατάστασή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ξέρω πως έχουμε καθυστερήσει. Είναι η κυρία Μακένης, αν ε, δεν κάνω λάθος με το όνομά σου. Σας παρακαλώ πολύ, για δύο-τρία λεπτά έχετε το λόγο. Εσείς εκπρε... εκπροσωπείτε το γραφείο της ΥΠΑ Αρμοστίας για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα είμαι όσο πιο σύντομη μπορώ. Σας, Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε σήμερα στη συνεδρίαση. Είναι μια πολύ χρήσιμη ένα χρήσιμο θέμα, όχι μόνο σε σχέση με την συγκεκριμένη κατάσταση στην Ιταλία, αλλά και γιατί η προσέγγιση της μετεγκατάστασης και των hot spot είναι αυτή που θα επιτρέψει ένα σωστό σύστημα να εγκαθιδρυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθήσει τη σωστή διαχείριση των χώρων προστασίας και της κατανομής ευθύνης. Είναι κρίσιμο λοιπόν αυτή η προσέγγιση για τα hot spot όπως εφαρμόζεται στην Ιταλία και το θέμα της μετακατάστασης να εφαρμοστούν πλήρως και ξέρω πως ανησυχούν πολύ όλοι πως μέχρι στιγμής μόνο 2.180 άτομα έχουν ε, μετακατασταθεί από την Ιταλία και από την Ελλάδα και από την Ιταλία μόνο 780. Ο στόχος που είχε η Κομισιόν ήταν 6.000 το μήνα. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ μακριά από το στόχο μας και θα θέλαμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Ονίδη αναφέρθηκε σε πολλές από τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και συμφωνούμε απόλυτα με την αξιολόγησή του και με τις συστάσεις που παρουσίασε για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Και υπάρχουν κάποιες επιπρόσθετες προκλήσεις, για παράδειγμα ο χρόνος απόκρισης από τα κράτη-μέλη που έχουν αναφέρει πως θα δεχθούν μεταγκαταστάσεις είναι υπερβολικός, δηλαδή σε σχέση με την Ιταλία υπάρχει το θέμα του screening για θέματα ασφάλειας και κάποια κράτη-μέλη επιμένουν να κάνουν και τη δική τους διαδικασία screening ασφάλειας, μια και, ε, και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι οι Ιταλικέ Αρχέ. Είδατε την έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από χτε, που λέει πω θέλουμε μια ε, ισορροπημένη ε, προσέγγιση που θα βοηθήσει αυτό το πρόβλημα να το ξεπεράσουμε. Επίση, χρειάζεται να παρουσιάσουμε την απαιτούμενη ε, βοήθεια στις Ιταλικές Αρχές και εμείς ως είπατε αρμοστία είμαστε επιτόπου αλλά χρειαζόμαστε ικανό αριθμό εμπειρογνώμων μέσω της ΕΑΣΟ και θα ήταν χρήσιμο αν τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατόν σε αυτή την πρόσκληση να έρθουν εμπειρογνώμονες από την ΕΑΣΟ και επίσης να επιτρέπουν στους εμπειρογνώμονες ΕΑΣΟ να παραμένουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι λίγο σύντομα ε, όταν αυτοί βρίσκονται επί τόπου. Τώρα, για το δυναμικό. Στα τέσσερα, ε, στα τέσσερα λειτουργικά hot spot ε, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω και χάρηκα που άξω τον κύριο Νίδρα μιλά για τα δύο επιπλέον hot spot που θα δημιουργηθούν. Χρειάζεται είναι απαραίτητο οι αφήξει στην Ιταλία να περάσουν από τα hot spot για να μπορούν όλοι να καταγράφονται σωστά. Το Μάιο είδαμε ότι το ποσοστό των ανθρώπων που πέρασαν από τα hot spot ήταν κάτω από το 45%. Θέλουμε να φτάσουμε στο στόχο του 100%. Ε, βέβαια όσοι ε, έφταναν τα ε, δακτυλοσκοπούνταν τουλάχιστον δηλαδή το 90%. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει πως οι διαδικασίες λειτουργούν. Να πω και δύο λόγια για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Θέλουμε οι ανισοδυνόδευτοι ανήλικοι να μετεγκατασταθούν, γιατί ξέρετε πως αποτελούν μια προτεραιότητα στην απόφαση του Συμβουλίου για τις μετεγκαταστάσεις και όλοι έχουν συμφωνήσει τα παιδιά αυτά να θεωρηθούν προτεραιότητα. Αυτό δεν συνέβη στην πράξη και αυτό για μια σειρά από λόγους. Υπάρχει περιορισμένος αριθμών χωρών που έχουν πει πως θα πάρουν ανήλικα παιδιά και θα πρέπει να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση που θα μας επιτρέψει πως, ε, να ληφθούν υπόψη βάσει του συμφέροντος των παιδιών αυτών και να βοηθηθούν με την όλη διαδικασία τα ανήλικα παιδιά. Και έχουμε προτείνει ε, πως θα πρέπει η διατάξεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τους ανήλικους θα μπορούσαν να βελτιωθούν και οι Ιταλικές αρχές μαζί με την Κομισιόν και άλλους εταίρους έχουν αυτή τη στιγμή ε, παρουσιάσει μία σειρά ε, στάνταρ πρακτικών που θα μπορούσαν όλοι να ακολουθούν. Θα πρέπει λοιπόν στους νέους και στους ανήλικους να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Είναι σημαντικό να το δούμε τώρα και όχι μόνο επειδή το 12% των αφήξεων είναι ανήλικοι, αλλά γιατί αυτό εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική του Κοινοβουλίου των Θεσμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πως προτεραιότητα δίνουμε στα παιδιά, το αφήνω εκεί και ό,τι ερώτηση έχετε με χαρά να απαντήσω. Ευχαριστώ συνάδελφε κύρια Μαγκένης Μαλό. Θα διαβάσω τον κατάλογο. Κοέλιο, Γκόμες, Πινέλη, Δίκστρομ, κύριος Αλαάχο, Σλέιν και Πουλιέζε. Πρέπει να κλείσω τον κατάλογο των αγορητών γιατί χρόνο δεν θα έχουμε και θα σας δώσω δύο λεπτά ανά άτομο. Κύριε Κοέλιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Φοβούμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι χειρότερη από ό,τι στην Ιταλία. Η ερώτησή μου είναι η εξής στην αρχή τα hot pot για τους περισσότερους από εμά έμοιαζαν να είναι καλή ιδέα. Το πρόβλημα όμω είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλαπλές δυσκολίες. Μερικά από αυτά τα αναφέρατε. Δυσκολία να ε, εξετάσουμε τις αιτήσει. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φτάνουν και δεν υπάρχουν πόροι. Δεν έχουμε τους ανθρώπινους πόρους για να καλύψουμε όλες τις απαραίτητες ανάγκες. Καθυστερούν λοιπόν πάρα πολύ στην πράξη. Και όχι μόνο οι δεσμεύσει των κρατών μελών καθυστερούν τι επιστροφέ. Διότι στη χώρα μου, την Πορτογαλία, που ήμασταν πρόθυμοι να αποδεχτούμε περισσότερου ανθρώπου, δεν μα έστειλαν πρόσφυγε. Διαθεσιμότητα υπάρχει, προθυμία υπάρχει, αλλά κανεί δεν έρχεται. Και μιλήσατε για συνόδευτου ανηλίκους ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα και μια από τι σοβαρότερε αρμοδιότητε των hot είναι να κάνει τον, τη σωστή ταυτοποίηση και να έχουμε περισσότερη ασφάλεια. Ξέρουμε ότι πολλά παιδιά και έφηβοι απέδρασαν αφού καταγράφηκαν. Είναι χιλιάδες. Οπότε το ερώτημα είναι μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε το μοντέλο των hot spot ή είναι απλώς ένα θέμα δυνατοτήτων. Τι δεν πάει καλά. Τι θα έπρεπε να κάνουμε καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή των φορέων και των κρατών μελών. Τι είδους πίεση πρέπει να ασκηθεί στα κράτη-μέλη. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα στην Ιταλία μπορεί να επιληθεί με δύο παραπάνω hot spot και δύο μόνο τέσσερα, και, με τέσσερα παραπάνω πλωτά Hotspot. Είναι θέμα δυνατοτήτων. Πρέπει να τα ξανασκεφτούμε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζίπελ, θέλετε το λόγο, όχι. Κυρία Γκόμερ. Ναι, και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε που αντιφάσκουν τελείως με όσα μας είχε πει ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς. Τι φοβερέ αυτές δηλώσεις ότι η ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας πηγαίνει καλά. Καλά πηγαίνει για να περιοριστούν οι αφήξει στην ε, Ελλάδα, αλλά τώρα έρχονται από την Ιταλία και την Αίγυπτο οι μετανάστες. Αυτό σημαίνει αύξηση αριθμού αφήξεων από την Αίγυπτο. Και βεβαίω αυτό έχει να κάνει και με την κατάσταση στην Αίγυπτο. Πλήρη έλλειψη ελέγχου ασφάλεια κλπ. Παρά τα τόσα πολλά που προσπάθησαν να κάνουν οι, ηγέτε, οι ηγέτες μας, οι, οι εταίροι μας και οι ομολογοί μας εκεί. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι οι λαθρέμποροι συνεχίζουν να βγάζουν λεφτά εις βάρος των ανθρώπων. Το είπατε. Είπατε ότι ο αριθμός των θυμάτων διπλασιάστηκε. Διπλασιάστηκε. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος Κοέλιο, Όντως, στην Πορτογαλία δεν έχουμε πρόβλημα να δεχτούμε μετανάστε. Δεν έχουμε απαγορεύσεις. Πέραν αυτών που είχατε από κάποια κάτι μέλη που επέβαλαν δικό του screening για δικού του λόγου ασφαλεία. Τι άλλε απαγορεύσει έχετε ακούσει. Διαλέγουν να βάζει το χρώμα των ανθρώπων, τη θρησκεία, τι πεπιθήσει του, αποκλείουν του νεαρού άντρε λόγου χάρη. Προτιμούν του ανηλίκου. Είναι σημαντικό για μας να γνωρίζουμε, ε, για να ξέρουμε αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση και θα εκτιμούσα πολύ μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόμες και τώρα κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον ε, κύριο Ονίδη για την παρουσίασή του. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτη. Μπορείτε να μου πείτε εσείς οι η ε, του UNHCR μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει κίνδυνο στα hot spot να μετατραπούν σε κέντρα κράτησης. Υπάρχει μια σαφέστατη καταγγελία από την ύπατη αρμοστία των προσφύγων προς αυτή την κατεύθυνση για την Ελλάδα και βάσει της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ίσως βεβαίως να ε, συμβεί κάτι τέτοιο και στην Ιταλία. Και το δεύτερο που ήθελα να ε, μου απαντήσετε είναι τα ε, πλωτά hot spot, αυτά που βρίσκονται στη θάλασσα. Με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα την πληροφορία αυτή ότι θα είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός δυνατών αρμοδιοτήτων που θα έχουν αυτά τα πλωτά hotspot. Διερωτώ με όμως, μήπως και αυτές οι αρμοδιότητες που αναφέρατε, όπως η προ-ταυτοποίηση, είναι ίσως υπερβολικά μήπως απλώς επιταχύνουν τις, τους επαναπατρισμούς να θυμίσω ότι υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της βάρο ε, βάρος της Ιταλίας για τη χρήση, την ενδεχόμενη χρήση που γίνεται των, σκαφών εκεί όπου πολύ σύντομα στηβάζονται, οι, πολύ γρήγορα μάλλον στηβάζονται οι μετανάστες και να πω ότι μόνο στην ξηρά μπορεί να λάβουν συνδρομή οι μετανάστες, να ε, έχουν γλωσσική εξυπηρέτηση και ακόμη και δικαίωμα στο ευεργέτημα παινίας. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη, κυρία Βίκστρομ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας, ειδικά να ευχαριστήσω θερμά για το γεγονός ότι υπογραμμίσατε τη σημασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, όχι μόνο στα hot spot στην Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα και αλλού. Συγκεκριμένα μιλώ για τα χιλιάδες παιδιά που εξαφανίζονται και εξαφανίζονται από τα hot spot και ε, ε, από όλα τα ραντάρ ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική στα hot spot στην Ιταλία έτσι ώστε να μην εξαφανίζονται και να μην μπαίνουν μέσα στα άγρια δίκτυα της Ευρώπης. Ε, είναι πολύ μεγάλη διάρκεια των εξαφανίσεων, πολλές, ε, πολλοί μήνες. Ε, όταν μιλώ με τις ΜΚΟ, για να το πω έτσι πιο ελαφριά, συνήθως επικρίνουν την προσέγγιση. Ε, ποια είναι αυτή. Συνήθως ενθαρρύνονται οι πρόσφυγες να φύγουν, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να φύγουν. Είναι ένα ακριβό ταξίδι αν θέλει κανείς να το κάνει σε τακτική βάση. Και ξέρουμε ότι περισσότεροι από όσου βρίσκονται στην Αφρική είναι από την υποσαχάριο Αφρική. Αν κανείς λοιπόν θέλει να αγοράσει ένα κανονικό εισιτήριο, ε, είναι ακριβό. Και επίσης δεν υπάρχει και μεταγκατάσταση. Δεν λειτουργεί βάση του ε, σχεδίου με το οποίο ε, έχουμε συμφωνήσει και φυσικά ούτε, ούτε και απέλαση. Ε, να, ακόμα και αν θέλει κανείς να φύγει δεν μπορεί. Ο απαναπατρισμός λοιπόν δεν λειτουργεί. Πρέπει επίσης να αυξήσουμε ε, την αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους αυτούς εντός των hot στην Ιταλία κάθε φορά τους αναφέρουν ως κλαντεστίνοι που σημαίνει χωρίς έγγραφα αν το καταλαβαίνω σωστά. Μπορείτε λίγο να μας πείτε κάποια πράγματα για την ε, κοινή γνώμη στην Ιταλία. Πώς τους βλέπει αυτούς τους ανθρώπους και ποιο είναι το επόμενο στάδιο στην προσέγγιση που έχετε για τα συνόδευτα ανήλικα. Ευχαριστώ κυρία Σλέιν. Ευχαριστώ. Έχει δίκιο ο συνάδελφο ε, Βίξτρομ για να ξεκινήσω. Κλαντεστίνη, λαθρέοι, είναι όρο που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Μπορούμε να μιλάμε για μετανάστε χωρί έγγραφα, αλλά πρόκειται πραγματικά για επινόηση ιταλική και τελείω ε, όργανο χειραγώγηση. Ε, είσαστε πολύ αισιόδοξοι για την λειτουργία των χώρων που στην Ιταλία. Εγώ επισκέφτηκα δύο τουλάχιστον και με άλλο συνάδελφο επισκεφτήκαμε και αυτό το ποτσάλο και να σας αναφέρω μερικές ειδήσει που δεν φτάνουν πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο, ακτιβιστών πολλές φορές που προσπαθούν να βελτιώσουν ακριβώς τη ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτά τα hot spot ε, και κάποιες φορές καλύπτοντας και τις ελλείψεις των κρατικών υπηρεσιών. Στη Λαμπεντούζα, λόγου χάρη. Το συζητήσαμε πολύ και με τη Δήμαρχο εκεί. Το νησί δεν προσφέρεται για να γίνει τόπος κράτησης ε, μακράς διαρκείας αυτών των ανθρώπων. Είναι γενναιόδοροι κάτοικοι του του νησιού αυτού δίνουν φιλοξενία και βοήθεια σε μια πρώτη φάση, αλλά πρέπει σε 48 ώρες τα άτομα αυτά να πάνε σε εγκαταστάσεις πιο κατάλληλες στην ε, ξηρά, στην υπόλοιπη χώρα. Ε, κατά τα άλλα δεν μπόρεσα να συναντήσω ε, υπαλλήλους της ΕΑΖΟ και της Frontex. Ίσως να ήμουν ατυχής εγώ γιατί δεν ήταν εκεί εκείνη τη μέρα. Αλλά οι επανακαταστάσεις, όπως λέγεται, πρέπει, ναι, πρέπει να φύγουν. Τα άτομα αυτά όμως πρέπει να έχουν μια σαφή προοπτική για το μέλλον τους. Ιδάλλως, προφανώς, θα είναι καχύποπτοι για να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα επανακατάστασης. Και ακόμα και να δεχτούν και την ταυτοποίηση. Τώρα, στο hot spot του Τάραντα, οι αρχές μας έδειξαν τις διαδικασίες και τις εγκαταστάσεις, μας είπαν πώς ε, πληροφορούνται οι μετανάστες σε διάφορες γλώσσες, μας έδειξαν τα έντυπα και τα άτομα απ' έξω μας είπαν ότι δεν είχαν πάρει τίποτα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς στην πράξη γίνονται αυτές οι συζητήσεις ενημέρωσης. Πολλές φορές στις εγκαταστάσεις υπήρχαν ανήλικοι και υπάρχουν κυβερνητικέ οργανώσεις που παραπονούνται και ακτιβιστές που παραπονούνται ότι κάποιες εθνικότητες συγκεκριμένα ε, δίδεται αμέσως το λεγόμενο λεσέπασε μέσα σε 7 ε, μέρες χωρίς όμως να τους έχουν γνωστοποιηθεί τα δικαιώματα που διαθέτουν οι άνθρωποι αυτοί όπως λόγω χάρη το δικαίωμα στη διεθνή προστασία και πάλι δεν υπήρχαν εκεί υπάλληλοι τη ΕΑΖΟ και τη Frontex και επίσης δεν είναι σαφέ με τι ασχολείται η ΕΑΖΟ και με τι Frontex η ΕΑΖΟ ασχολείται με τις πληροφορίες για τις μετακαταστάσεις η Frontex αναρωτιόμαστε τι κάνει ακόμα στα hot spot της Ιταλίας και ένα άλλο σημαντικό θέμα διάρκεια παραμονής όχι παραπάνω από 72 ώρε. Όμω πολλοί άνθρωποι μα λένε ότι μένουν εκεί μέχρι και μία εβδομάδα χωρί να ξέρουν τι να περιμένουν. Και τελευταία παρατηρήση, με συγχωρείτε για την ε, καθυστερήση, το hot, το hot spot του Ποτσάλιο. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ανήλικοι. Και μάλιστα μα είπαν ότι κυκλοφορούν ξυπόλοιτοι. Του είδαμε. Ε, χωρί ρούχα, που θα, τα απαραίτητα τουλάχιστον ρούχα, με λίγο, λίγα τρόφιμα. Μιλάμε για ζωέ που βρίσκονται σε αναστολή, σε κατάσταση εκκρεμότητα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ε, ευχαριστούμε, αλλά πρέπει να σεβόμαστε το χρόνο, συνάδελφοι. Ε, ακόμη δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο, ο κύριος Αλάχο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα που έχει αλλάξει η πίεση και έχει φύγει από την ελληνοτουρκική μεθόριο και έχει περάσει στην κεντρική Μεσόγειο, πώς επηρεάστηκαν οι αμοιβέ που ζητούν οι, οι λαθρέμποροι για να περάσουν ανθρώπους. Γιατί είπατε πως βάζουν όλο και περισσότερο στις βάρκες και οι βάρκες είναι όλο και σε χειροτερή κατάσταση. Ε, έχετε εντοπίσει ε, κάποιο λόγο γι' αυτό εκτός από το αυξανόμενο κέρδος. Και επίση, ποιο είναι ο προβλεπόμενο αριθμό αφήξεων για τη Μεσόγειο φέτο ή τουλάχιστον τι προβλέπετε μέχρι τα τέλη τη χρονιά. Έχετε κάποιε τάσει για τι υπηκότητε των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στα hot spot. Επίση, πόσοι από αυτού είναι από χώρε ε, ε, για τις οποίες μάλλον δεν θα χορηγηθεί διεθνή προστασία για παράδειγμα, είναι λιγότεροι αυτοί που θα είναι από τη Συρία από ό,τι ακούω. Ευχαριστώ πολύ. τελευταίο, είναι ο κύριος Πουλιέζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Νίδη για την παρουσίασή του, η οποία ήταν φοβερά διεξοδική και λεπτομερής. Νομίζω προκύπτει ότι συνολικά η κατάσταση των χώρων στην Ιταλία είναι θετική. Εν μέρη Διαφωνώ σε σχέση με αυτό που πει Ταλίδα συνάδελφο. Θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση σίγουρα. Αλλά εδώ πραγματικά καταγράφουμε ούτω ή άλλω την προσοχή που δίνει η Ιταλική κυβέρνηση στη λειτουργία του. Η συμφωνία με την Τουρκία όντω ε, μπλόκαρε την εδώ των Βαλκανίων και αναφέρεται και κάποια στατιστικά δεδομένα. 87% ε, των αναχωρήσεων ως σήμερα από τη Λιβύη, 12% ε, ξεκινά τελικά από την Αίγυπτο. Ε, και είδαμε να υπάρχει αύξηση των αναχωρήσεων από την Αίγυπτο. Είπατε επίσης ότι συγκυριακά οι εθνικότητες παραμένουν περίπου ίδιες με αυτές που είχαμε προηγουμένως. Ε, λίγους Σύρους, λίγους Ερυθρέους, λίγους Πακιστανούς και Αφγανούς. Όμως η αύξηση της μετακίνησης με σημείο αναχώρησης από την Αίγυπτο Αίγυπτο, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερο ποσοστό αυτό των εθνικοτήτων. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν τι γίνεται του τελευταίου μήνε μετά την εφαρμογή τη συμφωνία με την Τουρκία. Και για να κλείσω, ε, το είπατε νομίζω, είναι αποτυχημένη ω τώρα η λειτουργία του συστήματο τη επαναγκατάσταση και του, ε, των ε, επανεπατρισμών. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Ω σήμερα μόνο 787 είναι οι μετανάστες που έγιναν δεκτοί σε άλλα κράτη ξεκινώντας από την Ιταλία και 503 από την Ελλάδα. Ε, αν αυτό ήταν ο αρχικό μα στόχο, δεν νομίζω. Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ ακόμα από, το 2000, από του 2000. Όμω πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια από τα κράτη-μέλη και να, υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύστημα αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Πολιέζε. Και τώρα κύριε Ονίδη, έχετε το λόγο για τι απαντήσει σα και τα σχόλιά σα. Και σε εσά, κυρία μου, ο κύριο Ονίδη πρώτο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για αυτές τις τόσο πολύτιμες παρατηρήσεις και πάλι σε επίπεδο δεν θα προσπαθούσα να κάνω καμία πρόβλεψη για το συνολικό αριθμό που θα έχουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά από την περσινή χρονιά. Δηλαδή ούτε στον αριθμό, ούτε ε, στη χώρα προέλευσης και καμία διαφορά ε, και στα σημεία από τα οποία αποπλέουν. Οι δύο διαφορές που υπογράμμισα είναι ότι πρώτος έχουμε μία πρόσφατη τάση αύξηση από την Αίγυπτο, κάτι το οποίο μας ανησυχεί και αυτή τη στιγμή τρέχουν και κάποιες συζητήσεις με τις Αιγυπτιακές αρχές για να δούμε εάν υπάρχει κάποια δυναμία στο σύστημα εκεί. Και επίσης έχουμε μια άλλη διαφορά που μάλλον έχει να κάνει με την μεγαλύτερη απληστία των τράφικερς, που έχει να κάνει με τον ε, μεγαλύτερο αριθμό θνησιμότητας σε σχέση με την περσινή χρονιά μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας. Οι κατηγορίες ε, ε, μεταναστών που έρχονται από την Κεντρική Μεσόγειο και, την και τα Ανατολικά Βαλκάνια είναι ακριβώς όπως ήταν. Δηλαδή, στα Βαλκάνια είχαμε πολύ περισσότερους οικονομικούς μετανάστες από ότι ε, τούντες άσυλο. Για τα hotspot Νομίζω ότι δεν έχουν ούτε ένα χρόνο ζωής και δεν θα έλεγα πως δεν λειτουργούν τα hot spot, θα έλεγα πως αποτελούν μια καταπληκτική επιτυχία όπου όμως υπάρχει και, μεγάλος, και μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και σίγουρα κάποια στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα, ίσως ένα χρόνο μετά το, την έναρξη λειτουργίας αυτών για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και κυρίως μετά τη θερινή περίοδο. Να δούμε δηλαδή τι είδου βελτιώσεις μπορούμε να εισάγουμε στο σύστημα. Δεν πιστεύω πως τα hot spots στην Ιταλία ε, είναι άδεια σε επίπεδο αξιωματούχων ΕΑΖΟ και Frontex. Ίσως ήταν μια πολύ ατυχή σύμπτωση και αντίθετα θα έλεγα πως αυτό που είπε η συνάδελφος στην ύπατη αρμοστία είναι αλήθεια. Απλώς δεν έχουμε αρκετά άτομα από αυτά τα οποία είχαν δεσμευτεί τα κράτη τα οποία θα στείλουν. Δηλαδή επαγγελματίες οι οποίοι θα συνοδεύσουν αυτή την τάση και μια ενδεχόμενη αύξηση αλλά υπάρχει κόσμος επί τόπου. Και εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε τρία άτομα τα οποία ε, ε, με ενεργό τρόπο ε, αυτά τα hot spot για να είμαστε σίγουροι πως μπορούμε σε γρήγορο χρόνο να ανταποκριθούμε και να προτείνουμε αλλαγές αν χρειάζονται. Το κρίσιμο σημείο δυναμίας που βλέπει κανείς στα hot spot δεν είναι η λειτουργία του hot spot, αλλά το γεγονός πως οι λειτουργίες που κάνουν εκεί είναι περιορισμένες. Δηλαδή, καταγραφή, ταυτοποίηση και συμβουλή. Συμβουλεύονται από την ΕΑΣΟ για τα δικαιώματά τους οι νεοφυχθέντες. Όλα αυτά όμως μπορούν να υποκαταστήσουν την πραγματική στέγαση, αποκατάσταση, εκπαίδευση και κυρίως όταν μιλάμε για ανήλικους. Άρα λοιπόν αυτό είναι άλλο κομμάτι της διαδικασίας και εκεί ίσως εξετάζοντας την μελλοντική εξέλιξη των hot spot μπορεί συλλογικά να δούμε πως θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να το προσθέσουμε αυτό το στοιχείο έτσι ώστε και σε αυτά να έχουμε κάποιες παραπάνω δικλείδες ασφαλείας. Τώρα για την κατάσταση στην Ιταλία θα πρέπει να ε, απευθύνω εύσημα στις Ιταλικές αρχές γιατί σε επίπεδο δυναμικού και σε συνθήκες και δυναμικού υποδοχής περνάμε από τις 125.000 θέσεις σήμερα στις 200.000 θέσεις στα τέλη του καλοκαιριού. Μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε έτοιμοι, έχουμε τα χρήματα, αλλά πρέπει, και εδώ επιστρέφω στο θέμα των ασυνόδευτων ανήλικων, πρέπει να έχουμε ασφαλείς που είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα και κρίσιμο για να καταφέρουμε τουλάχιστον να βοηθήσουμε να καταφύγουν κάπου αυτοί οι ανήλικοι, να τους κατευθύνουμε, να τους προσφέρουμε παιδεία, όσο περιμένουν κάποια πιο βιώσιμη λύση για το μέλλον τους. Ευχαριστώ η κυρία Μαγκίνης. Ευχαριστώ Πρόεδρε να επανέλθω σε κάποια από τα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί, γιατί υπόθηκε ε, τι θα μπορούσε να γίνει για να λειτουργήσει καλύτερα η διαδικασία μετακατάσταση. Ήδη έχει αναφέρει ο κύριο Ονίδη κάποια πράγματα. Οι ε, διαδικασίε διαδικασίες ε, αποφασίστηκαν τον Μάιο σχετικά με τα hot spot στην Ιταλία. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και οργανισμών. Η ε, καλή λειτουργία των διαδικασιών είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει στοχοθετημένη ε, εξέλιξη για όλα όσα γινόνται σχετικά με τους ε, ε, ασυνόδευτους ανήλικους. Εμείς ε, αυτό που λέμε στην αρμοστία είναι ότι πρέπει να δρούμε πάντα με γνώμονα την προστασία των παιδιών και όχι τις διοικητικές διαδικασίες και αυτές τις ε, ε, τυπικές διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν εξ αρχής ε, σε πρώιμο στάδιο να διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν για αυτά τα παιδιά ότι έχουν σωστή ε, στέγαση και δεν εξαφανίζονται. Η μετεγκατάσταση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί οι ασυνόδευτοι και οι ευάλωτοι ε, που ε, ταυτοποιούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να έχουν κάποια σχέση με άλλα κράτη-μέλη ε, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δουβλίνου θα πρέπει να διευκολύνονται ως, ε, προς την επανένωσή τους με την οικογένειά τους. Αυτό όμως έχει αποδειχτεί δύσκολο γιατί κάποια κράτη μπορεί να έχουν πιο στοχοθετημένη προσέγγιση. αν μιλήσω για την Ελλάδα με την προ εγγραφή που ξεκίνησε η καταγραφή που ξεκίνησε τον Ιούνιο από τις ελληνικές αρχές μαζί με την ΕΑΣΟ και την ΥΠΑΤΗ για να μπορεί να γίνει η πρώιμη αυτή καταγραφή όσο πιο γρήγορα γίνεται ε, για όσο περισσότερους ανθρώπους γίνεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους που έχουν κολλήσει στην Ελλάδα και για να ταυτοποιήσουμε τους ε, ασυνόδευτους ανήλικους, τα εισεβάλλοντες ομάδες. Επίσης ε, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σύνδεση με τα άλλα κρατημέλη για να γίνουν αυτές οι μεταφορές. Αυτό να γίνει παράλληλα με το πρόγραμμα μετεγκατάσταση. Τέλος, ε, σχετικά με την ευρύτερη εικόνα, να πω ότι ένα από τα πράγματα που υποστηρίζαμε πάρα πολύ ήταν οι νομικέ οδοί. Δηλαδή, Αφήνοντας τη μετεγκατάσταση χρειάζονται και νομικές οδοί για τους ανθρώπους που δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Ευρώπη αλλά χρειάζονται μεσόδη για αυτούς τους ανθρώπους ε, που θέλουν να έρθουν εδώ. Υπάρχει, ε, όπως είπαμε, ένας μικρός αριθμός μετεγκαταστάσεων, αλλά και για την επανεγκατάσταση πάνω από 7.000 άτομα έχουμε. Αν θέλουμε να στείλουμε λοιπόν ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μπορεί να σκέφτονται να κάνουν ένα επικίνδυνο ε, ταξίδι είτε μέσω της κεντρικής οδού της Μεσογείου είτε από, την, από το Αιγαίο, αν θέλουμε να τους πούμε ότι υπάρχει εναλλακτική πρέπει να βρούμε κάποια αξιόπιστη οδό. Ε, είναι η νόμιμη οδός ε, η οποία όμως ε, θα πρέπει να ε, προβλέπει για μεγαλύτερα ποσοστά επανεγκατάσταση. Είπαμε πρόσφατα, ας πούμε, ότι θα θέλαμε το 10% των Σύριων να μπορούν να μπουν ε, σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, τα ανθρωπιστικά προγράμματα στην Τουρκία πρέπει να λειτουργούν, αλλά και από άλλες χώρες, από το Λίβανο και από την Ιορδανία, για παράδειγμα, πρέπει να έχουμε σωστή επανεγκατάσταση. Δεν πρέπει η Ιταλία και η Ελλάδα να φεθούν μόνες τους ε, να αντιμετωπίσουν αυτή την πίεση. Πρέπει όλοι να προωθήσουμε αυτή την νόμιμη οδό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μακγένης. Ευχαριστούμε κύριε Ονίδη. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Στις 4 Μαΐου 2016 η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο 3. Η πρόταση είναι το κεντρικό ε, σημείο του πρώτου πακέτου μέτρων ε, για την μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Η μεταρρύθμιση του συστήματος αυτού στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που έγιναν ε, εμφανείς κατά την τρέχουσα κρίση προσφύγων. Η πρόταση ε, άπτεται δύο προηγούμενων προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον λεγόμενο μηχανισμό ε, για την κρίση, σε περίπτωση κρίσης για τον οποίο ήταν ο κ. Κίρκοπ καθώς και την, τροποποίηση του κανονισμού του Βλήνου 3 ό,τι αφορά τον εντοπισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, δηλαδή ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων, για την οποία συγγέντρια ήταν η κυρία Βίξτρομ. Στις αρχές της φετινής χρονιάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις πολιτικές ομάδες για να μάθει τις απόψεις τους σε σχέση με, με τη μεταρρύθμιση του συστήματος Δουβλίνου και βάσει της ανακοίνωσης της 6 Απριλίου ε, καθόρισε δύο δυνατές για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε τον κύριο Μουσέλ, ε, Διευθυντή για τη Μετανάστευση και την Προστασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ο οποίο θα μα παρουσιάσει την πρόταση. Κύριε Μουσέλ, έχετε το λόγο. Merci, Madame la Présidente. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σα ε, παρουσίασε, όπω ξέρετε, πριν από λίγου μήνε την πρότασή τη για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Είναι μέρο του πρώτου κύματο νομοθετικών προτάσεων που υπευλήθησαν με σκοπό να μεταρρυθμίσουμε τελείω το Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου. Βεβαίω, η πρόταση περί Δουβλίνου είναι μια από τι πλέον αμφιλεγόμενε, είναι πολιτικά περίπλοκη, αλλά είναι και θεμελιώδου σημασία για τι αλλαγέ που χρειαζόμαστε ω προ το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Γνωρίζουμε όλοι ότι το να διατηρήσουμε το status quo όσο έχει δεν είναι επιλογή. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την περσινή κρίση ε, όπως συνέβη στην Ιταλία και στην Ελλάδα, μεμονωμένα, χωρίς ένα κοινό σύστημα. Έχουμε ένα διτό στόχο λοιπόν στη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. Ο πρώτος είναι οι κανόνες του Δουβλίνου να γίνουν αποτελεσματικότεροι και ο επόμενος είναι να προσθέσουμε όσα ε, ζητούνται από καιρό από το Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή ένα στοιχείο αλληλεγγύης, ένα παράγοντα αλληλεγγύης και δικαιοσύνης στο όλο σύστημα. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη ε, δεν μπορούν ε, να επομίζονται όλη την πίεση ενός κοινού συστήματος ε, μεμονωμένα. Να αναπτύξω τα δύο τώρα σκέλη. Πρώτα απ' όλα η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Θα πρέπει πιο σύντομα να αποστέλλονται οι αιτήσεις μεταφορές, να γίνονται δεκτές απαντήσεις και να γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα στους ετούντες άσυλο. Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει δυνατότητα για μετατόπιση αρμοδιοτήτων ε, και ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Αυτό προκαλεί τι δευτερογενεί και τριτογενεί μετακινήσει. Στο μέλλον, όταν ένα κράτο μέλο έχει εντοπιστεί ω υπεύθυνο, δεν θα μπορεί να ε, αναστείλει τι ευθύνε του. Να μην αναλάβει αυτέ τι ευθύνε. Ε, Επίσης θα πρέπει να ε, αποθαρρυνθούν περισσότερο οι, σε δεύτερη φάση κινήσεις με σαφείς ευθύνες για τους ετούντες άσυλο όπως το καθήκον να παραμείνουν στο κράτος που εξετάζει την αίτησή τους και να λάβ, εφόσον λαμβάνουν ουσιαστικά ωφελήματα από τον κράτος αυτό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δευτερογενείς όπως λέγονται μετακινήσεις εάν θέλουμε να είναι δίκαιο και αδηλέγγυο το σύστημα πρέπει να αποφύγουμε ή μετανάστες να παίζουν τους κανόνες του συστήματος και να καταστρέφεται το στοιχείο της αλληλεγγύης με δευτερογενείς μετακινήσεις. Να έρθω τώρα στο μηχανισμό αλληλεγγύης. Πραγματικά ε, έχει ονομαστεί διορθωτικός αυτός ο μηχανισμός. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει αυτόματος υπολογισμός του αριθμού ετούντων άσυλο που θα πρέπει να είναι δίκαιος στο όλο σύστημα. Θα βασίζεται σε δύο κριτήρια, δύο απλά κριτήρια, γιατί αποφασίσαμε να είμαστε απλοί και λιτοί, ε, με κάποια κριτήρια αναφοράς, όπως το μέγεθος της χώρας, ο πληθυσμός της και το ΑΕΠ της. Μέγεθος, πληθυσμός και ΑΕΠ. Αυτά θα είναι τα δύο βασικά κριτήρια. Για να καθορίσουμε ποιος είναι ο δίκαιος αριθμός των τον άσυλο πρέπει να παραλάβει. Το σύστημα θα υπολογίζει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των αιτήσεων και θα τις εξετάζει. Όταν ξεπεράσει καλής ε, την κλίδα αναφοράς, 150%, τότε θα θεωρούμε ότι θα υπάρχει δυσανάλογο βάρος και θα υπάρχει μετατόπιση του 50%, θα είναι μια άλλη κλίδα αυτή, ώστε να ισχύει το σύστημα παρέκκλησης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει και τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν ε, μετακατασταθεί από κάτι μέλη. Δηλαδή θα ενσωματώσουμε και το στοιχείο της μετακατάστασης ώστε τα κράτη-μέλη να αναγκαστούν να αναπτύξουν νόμιμες οδούς προς την Ευρώπη. Όπως μας είπε μόλις προηγουμένως η εκπρόσωπος από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία. Είναι σημαντικό να υπάρξει και αυτή η διάσταση. Ένα από τα στοιχεία που είναι αμφιλεγόμενο και το οποίο γνωρίζω καλά ε, είναι να υπάρχει δυνατότητα να μην συμμετέχει κανείς στο σύστημα επανακατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μία αλληλέγγυα συνεισφορά 250.000 ευρώ ανά μετανάστη που θα αποστέλλεται στο κατός μέλος και το οποίο θα έχει να κάνει με τη μία ανάληψη ευθυνών. Αυτός είναι ένας τρόπος για να επιτρέψουμε κάποια ευελιξία σε, σε κάποια μέλη. Όμως το ποσό που προβλέψαμε είναι αρκετά υψηλό. Οπότε ελπίζουμε ότι δεν θα ανατρέχουν σε αυτή τη δυνατότητα. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή σας, τουλάχιστον κάποια μέλη της Επιτροπής σας, θα προτιμούσαν τη δεύτερη επιλογή. Την δεύτερη επιλογή που προτείνει η ανακοίνωση και που πρότεινε η Πρόεδρό σας. Δηλαδή, να απαλλαγούμε από τα γεωγραφικά κριτήρια, να τα καταργήσουμε, τα κριτήρια πρώτη εισόδου των μεταναστών. Όμως ακούσαμε όλους τους ενδιαφερομένους και θεωρούμε ότι αυτό που προτείνουμε έχει πιθανότητες στη συναπόφαση να περάσει. Δεν υπάρχει λόγος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, η οποία να είναι πολύ όμορφη στο χαρτί, και να είναι ελκυστική, αλλά να μην πάει πουθενά στη συναπόφαση. Θέλουμε αυτό που θα θέσουμε επιτάπητος να φτάσει κάπου και στο, στο επίπεδο του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρξουν κριτήρια νόμιμης εισόδου, αλλά και αποτρεπτικά κίνητρα για να ελεγχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος με αυτά τα τρία νέα κριτήρια που θεσπίσαμε. Επίσης, δεν λάβαμε υπόψη τις προτιμήσεις των ετούντων. Δεν θα κοιτάζουμε πού θέλει να πάνε οι ετούντες άσυλο. Θέλουν να πάνε στη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πολωνία. Δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Διότι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε είναι ένα σύστημα ευρωπαϊκό για το άσυλο. Αναζητούμε, μάλλον αν ζητά κανείς προστασία στην Ευρώπη, δεν μπορεί να ζητά την προστασία σε ένα συγκεκριμένο κράτο μέλο, δεν μπορεί να επιλέγει και να του αρέσει ένα κράτο μέλο περισσότερο από ένα άλλο. Βεβαίω, μπορεί κάποιο να απαντήσει ναι, αλλά οι μετανάστε έχουν και κάποιε γλωσσικέ ικανότητε. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτέ. Κάποιοι έχουν συγκεκριμένα προσόντα. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αποφασίσαμε να μην το κάνουμε, διότι θέλουμε ένα σύστημα γρήγορο, αποτελεσματικό που να δουλεύει. Αν αρχίσουμε να προσθέτουμε και άλλα κριτήρια, το σύστημα θα γίνει φοβερά περίπλοκο και δεν θα είναι εύχριστο. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Όταν έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, γρήγορα να παρακαθίστανται. Ένα από τα κριτήρια που αλλάξαμε είναι το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης. Προσθέσαμε τα αδέρφια στον ορισμό της οικογένειας, καθώς και τις οικογένειες σε διέλευση. Ε, πολλές φορές κάποιοι είναι χωρισμένοι ε, για χρόνια, μήνες, μέρες ε, πρέπει να τους επιτρέπουμε να επανενωθούν κατά τη διέλευση. Το σύστημα του Δουβλίνου είχε πολύ ε, περιοριστικό ορισμό της οικογένειας. Τώρα έχουμε διευρύνει τον ορισμό της οικογένειας στο νέο σύστημα, στην πρότασή μας, για να καταπολεμήσουμε και τις δευτερογενείς, όπως λέγονται, μετακινήσεις. Διότι είναι λογικό ο μετανάστε να πάει εκεί που είναι η υπόλοιπη οικογένειά του και να μην είναι χωρισμένο από αυτήν. Να αποφύγουμε λοιπόν πίεση για δεύτερε μετακινήσει. Και το τελευταίο που θέλω να εντοπίσω είναι ότι αυτή είναι μια πρόταση από πολλέ. Εάν θέλουμε όμω να λειτουργήσει το σύστημα του Δουβλίνου, θα πρέπει να αναζητήσουμε την συμφωνία των 100 μελών και ω προ του όρου υποδοχή και ω προ τα ποσοστά αναγνώριση. Εάν ένας Αφγανός υποβάλλει αίτηση στο, στην Ιταλία θα πρέπει να έχει τις ίδιες πιθανότητες να περάσει η αίτησή του όπως αν την είχε υποβάλει στην ε, ε, Σουηδία ή τη Λετωνία. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Και αυτό θα το συμπληρώσουμε με τις υπόλοιπες προτάσεις μας. Δείτε το ως μέρος ενός πακέτου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπληρώσει το πακέτο και θα πίνει και άλλες ε, αναθεωρήσεις για την οδηγία όρων υποδοχής, για την οδηγία των προσόντων και για την οδηγία της ε, εξετάσεις των αιτήσεων ασύλου. Θα έρθουν εν αυτό το χρόνο και αυτές προτάσεις στα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μουσέλ. Και τώρα η κυρία Βίξτρομα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς να στραφώ στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Μισελ, και να τον ευχαριστήσω για την παρουσίαση και όλους ε, τους συναδέλφους που μου επέτρεψαν να μπορέσω να εργαστώ επί αυτού του πολύ σημαντικού θέματος. Όταν πριν από τρία χρόνια είχαμε το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, ε, οι περισσότεροι από εμά θεωρούσαμε ότι είχαμε θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο στην πράξη θα λειτουργεί για τους ετούντες άσυλο και για τα θεσμικά όργανα αλλά και τα κράτη-μέλη σε όλη την Ευρώπη υπήρξαν Πολλές φορές όμως ε, που η ομάδα του Κοινοβουλίου θα ήθελε να είχε κάποια διαφορετική προσέγγιση. Θεωρούσαμε όμως όλοι ότι είχαμε θέσει τα θεμέλια για ένα βιώσιμο σύστημα ασύλου που θα λειτουργούσε περισσότερο από ό,τι λειτουργήσε, δύο χρόνια δηλαδή. Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι το σύστημα κατέρευσε δεν μπορεί να δώσει πρόσβαση σε μια δίκαιη διαδικασία για τους ετούντες άσυλο, δεν δίνει στις αρχές των κρατών μελών τα εργαλεία που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτή τη συνεχή κατάσταση με τις συνεχείς αφήξεις τεραστίων αριθμών προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, επίσης ε, που έχει πληγεί πάνω απ' όλα είναι η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ξενοφοβικές ομάδες ε, να κερδίζουν σε δύναμη σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κάνει λοιπόν τώρα μία πολύ απρόσεκτη και τυχαία θέσπιση ατάκτως ηρημένων ε, μέτρων. Ε, για να, γι' αυτό χρειάζεται ένα σύστημα που θα μπορεί στην πράξη να λειτουργήσει. Μπορούμε λοιπόν τώρα να φτιάξουμε κάτι ε, που θα λειτουργήσει πολύ περισσότερο από ό,τι λειτουργήσε αυτό πάνω από δύο χρόνια. Είναι η πρόταση της Επιτροπής για το Δουβλίνο, την Eurodac, το ΕΑΖΟ και τώρα περιμένουμε και τις προτάσεις ε, για τα υπόλοιπα θέματα που σχετίζονται με το άσυλο, ε, όπως είναι η οδηγία για τα προσόντα, για την επανεγκατάσταση και ούτω καθεξής. Ε, τα στοιχεία αυτά αλληλοσυνδέονται. Είναι δύσκολο να δοθεί μία γνωμοδότηση για το σύστημα που προτείνει η Κομισιόν πριν τα δούμε όλα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να συνεργαστούμε στενά σε αυτή την Επιτροπή οι διάφορες ομάδες και οι συγητές επί των διαφόρων θεμάτων για να διασφαλίσουμε ότι θα δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα που θα έχει μία συνοχή θα πρέπει οι νομικέ πράξεις να αναθεωρηθούν με ένα βιώσιμο τρόπο όσον αφορά στον κανονισμό του Δουβλίνου που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Ε, εγκρίθηκε μια σειρά από ε, βασικές κατευθυντήριες αρχές ε, πριν από μερικές εβδομάδες με την έκθεση για τη μετανάστευση. Αυτές οι αρχές μπορώ να σας το εξασφαλίσω θα καθοδηγούν εμένα όταν ε, ε, σκέφτομαι το θέμα του κανονισμού του Δουβλίνου. Να πω ποια είναι τα κριτήρια που θεωρώ ότι πρέπει να πληρούνται πάνω απ' όλα. Πρώτον και κυριότερον, όποιο σύστημα και αν συμφωνήσουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λειτουργεί στην πραγματικότητα, στο πεδίο. Τα ευχολόγια πρέπει να σταματήσουν να τελειώνουμε με αυτά, γιατί οι σε άσυλο, οι πολίτες της Ευρώπης αξίζουν από εμάς ε, τους πολιτικούς ε, να τους δώσουμε ένα σύστημα ανθεκτικό που θα λειτουργήσει και να διασφαλίσουμε ότι όσοι έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα στην Ευρώπη. Δεύτερον, για να λειτουργήσει το σύστημα και να προχωρήσει σωστά, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών όσον αφορά στην υποδοχή των ετούντων άσυλο στα διάφορα κράτη-μέλη. Αν ε, μερικά μόνο κράτη παραμείνουν ε, στο προσκήνιο και μόνο αυτά αναλαμβάνουν την ευθύνη, το σύστημα θα ξανακαταρρεύσει. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το σύστημα ε, της ε, δίκαιης κατανομής ευθυνών δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις και δεν μπορούμε να τις ε, υποεκτιμούμε. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό θα αποτύχουμε. Το τρίτο κριτήριο είναι το εξή. Θέλουμε ένα σύστημα που θα δημιουργεί θετικά κίνητρα και θα δημιουργεί εμπιστοσύνη. Οι ετούντες άσυλο που φτάνουν στις ακτές μας θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι το σύστημα της Ευρώπης θα τους δίνει πρόσβαση σε μια δίκαιη ακρόαση και θα τους δίνει προστασία εφόσον πληρούν τα κριτήρια για τη διεθνή προστασία. Τα κράτη-μέλη επίσης πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι κάθε μία ξεχωριστά από τις 28 χώρες της Ευρώπης θα έχει το κίνητρο να παίξει σωστά το ρόλο της και στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Τα κράτη-μέλη επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα άτομα που έχουν τύχει δίκαιες διαδικασίες και ε, δεν πληρούν τα κριτήρια για τη διεθνή προστασία θα επιστρέφονται με αξιοπρεπή τρόπο στις χώρες τους οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ε, και να πιστέψουν ότι η Ευρώπη θα σταθεί στο ύψος των ιδεοδών και των υποχρεώσεων της και ότι θα μπορούν οι ευρωπαϊκές χώρες να διαχειριστούν τις ροές των μεταναστών με έναν τρόπο σωστό που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης. Να σας ε, πω επίσης, να σας διαβεβαιώσω, ότι έχουμε ξεκινήσει μια εντατική εργασία με τους σκιώδεις. Έχουμε κάνει δύο συναντήσεις και έχουμε ε, προγραμματίσει μέχρι τις διακοπές του καλοκαιριού να συναντιόμαστε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Φιλόδοξο σχέδιο και τούτου λεχθέντος να μην σας δώσω την εντύπωση, δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι τα πράγματα θα τα ε, λύσουμε έτσι γρήγορα. Ε, γιατί χρειαζόμαστε χρόνο για να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Επίσης να πω ότι έχω συνεχείς ε, συναντήσεις με ΜΚΟ, διάφορους εμπλεκόμενους, διεθνείς ε, οργανισμούς και άλλους που έχουν εμπειρία στο πεδίο από το τρέχον σύστημα για να μπορέσω να έχω μια ιδέα σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση. Ταυτόχρονα ήδη έχω ξεκινήσει μια σειρά συναντήσεων με τα κράτη-μέλη που είναι μάλλον το πιο δύσκολο γιατί παρόλο που ε, η αφετηρία, η θέση από την οποία ξεκινά ε, το ε, Κοινοβούλιο μπορεί να αντιβαίνει με αυτά που θέλουν κάποια κράτη-μέλη. Στο τέλος θα πρέπει να βρούμε μια κοινή θέση. Επίσης, θα πρέπει να μπορέσουμε ο καθένας να σταματήσει να περιχαρακώνεται πίσω από τις θέσεις του και να μπορεί να παλέψει μαζί με τους υπόλοιπους για τον κοινό στόχο. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να σταματήσετε. Θα τελειώσω. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε ένα κοινό σύστημα ασύλου το οποίο θα πέσει στο τραπέζι και θα μπορούμε συνεχώς με επικοδομητικό τρόπο να προσπαθούμε να βρούμε μια λύση η οποία θα επαναφέρει την αξιοπιστία του συστήματος. Αυτό το οφείλουμε στους ετούντε άσυλο, σε όλους όσοι δουλεύουν για να μπορέσουν να δώσουν μια σωστή υποδοχή στους ε, πρόσφυγες στην Ευρώπη και σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Έχουμε δυστυχώς αποτύχει παταγωδός. Όμως αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί. Συνάδελφοι, να σας διαβεβαιώσω ότι η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε έχει επικοδομητικές και δημιουργικές ιδέες για να μπορέσουμε όλοι μαζί να βρούμε τις σωστές λύσεις. Είμαι πεπισμένη, όχι μόνο ότι μπορούμε, αλλά ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Δίκστρομ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε εδώ έξι σκιώδεις εισηγητές αλλά βλέπω στην αίθουσα να είναι μόνο η κυρία Σλάιν. Μήπως η κυρία Μέτσολα μπορεί να βρει κάποιον να παρουσιάσει τη δική της ε, έκθεση. Όχι. Κυρία Σλέιν, έχετε το λόγο. Ε, thanks, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ. Δεν αποτελεί μυστήριο για οποιονδήποτε το γεγονός ότι εμάς δεν μας ε, ικανοποίησε η προτινόμενη μεταρρύθμιση της συνθήκης του Δουβλίνου και είναι πολύ μακριά ότι ψηφίσαμε εμείς στη σχετική έκθεση. Μας ζητήσαν να ε, ο, ξεπεράσουμε την αρχή της χώρας πρώτης αύξησης με ένα αυτόματο μηχανισμό κατανομής ευθυνών ανάμεσα κράτη-μέλη και ζητήσαμε μια πραγματική κεντρική διαχείριση της διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, Έχουμε εδώ ένα διορθωτικό μηχανισμό εξισορρόπησης, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα ενεργοποιείται και πώς θα λειτουργεί. Το κριτήριο που ακολουθείται εδώ των 150% είναι καθαρά μαθηματικό και δεν λαμβάνει υπόψη το τι γίνεται με τις συνθήκες υποδοχής ε, κάποιων κρατών μελών που ήδη καταραίων. Επίσης, ο προσωρινός αποκλεισμός πώς λειτουργεί, ανανεώνεται ή θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αιτιολογήσουν αυτή την απόφαση με κάποιο τρόπο είναι πολύ δύσκολο να πιστεύουμε πως η οικονομική αλληλεγγύη θα επαρκεί. Γιατί με την ε, πρώτη χώρα άφηξης, ε, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, να έχουμε ακόμα μία δυσαναλογικότητα, γιατί χρειάζεται κάποιοι έλεγχοι που θα γίνονται στο πρώτο χώρο, στην πρώτη χώρα άφηξης, για το θέμα της ε, δυνατότητας αποδοχής του ατόμου αυτού, όπως επίσης και κάποιοι έλεγχοι για το προφίλ ασφάλειας του ατόμου για τις προτιμήσεις που αναφερθήκατε κι εσείς, το Κοινοβούλιο στο παρελθόν έχει υπογραμμίσει την ανάγκη λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις που εκφράζουν οι αιτούντες άσυλο. Και στην έκθεση Κέλλερ είχαμε κάτι τέτοιο πέρυσι. Πιστεύω πως είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε τη δευτερογενή μετακίνηση ε, και αν κατάλαβα καλά, ο τρόπος που τα κράτη-μέλη κατανομής αποφασίζονται ε, είναι ε, μία λαχιοφόρος αγορά Άρα λοιπόν αυτό ξεκινά από την αρχή πως κανένα κρατομέλος δεν επιθυμεί να κάνει αυτό που χρειάζεται. Δεν είναι κοινικό αυτό. Ίσως κάποια κράτη-μέλη θέλουν να κάνουν αυτό που πρέπει και ίσως θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Θα το πω για τελευταία φορά επειδή το θίξατε κι εσείς. Δεν νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εάν είχε προτείνει πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση, θα είχε χρειαστεί να κάνει πίσω. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, κάποιοι που θα την υποστήριζαν και στο Συμβούλιο. Και εδώ χάθηκε μια ευκαιρία. Οι κυβερνήσει που δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τη και δεν θέλουν να δείξουν αλληλεγγύη, να μην φανούν. Γιατί θα μπορούσαν πραγματικά ε, να τεθούν ενώπιον των πολιτικών του ευθυνών. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πολύ στενά για τη μεταρρύθμιση αυτή. Είναι εξαιρετική ομάδα που είναι διαθέσιμη και επικεφαλής της ομάδας η συνάδελφος Βίξτρομ είναι εξαιρετική στη δουλειά της. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε την πρόταση αυτή όσο πιο παρόμοια με αυτά τα οποία ζητήσαμε εδώ και πάρα πολλές φορές στο Κοινοβούλιο, όπου κανείς βέβαια δεν άκουσε τι λέγαμε με αρκετή προσοχή είναι επόμενο Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω, αγαπητοί συνάδελφοι. Και πρέπει να σας πω ότι εκ μέρου της συναδέλφου κυρία Μέτσολα θα ήθελα να σας πω πως Καταρχήν πρέπει να απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία προσπάθησε να βρει κάποιες λύσεις για την κατάσταση αυτή. Ξέρετε πως χρειάζεται να είναι πολύ δραστήρια και για τα έγγραφα αυτά τα οποία προτείνονται και όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι ευδρομιγραμματίζονται παραπάνω με την πραγματικότητα που έχουμε. Αυτά ως κυρία Μέτσολα. Τώρα προσωπικές απόψεις. Έχω και μια ερώτηση να σας απευθύνω. Και είναι κάτι το οποίο αναρωτήθηκα όταν σας άκουσα να κάνετε την παρουσίασή σας. Μας είπατε, και να είμαι πιο ειλικρινής, 7 σύντομες ερωτήσεις θα σας κάνω. Οπότε ελπίζω να μην με σταματήσει η Πρόεδρος. Καταρχήν, ποιος είναι ο υπεύθυνο για το κόστος μεταφοράς. Είναι το κράτος μέλος από το οποίο ξεκίνησε η μεταφορά ή το κράτος μέλος όπου μεταφέρεται το άτομο αυτό. Γιατί αν το άτομο συμπεριφερθεί άσχημα, δείξει βίαιη συμπεριφορά, ε, κάνει κάποιο, ε, διαπράξει κάποιο έγκλημα ή πού θα δικαστούν. Δεύτερον, Ποιο θα πληρώσει για την ίδια τη μεταφορά. Γιατί το άτομο αυτό θα συνοδεύεται με κάποιο τρόπο, ε, ίσως θα πάρει αεροπλάνο ή θα πάρει αυτοκίνητο. Μετά, πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτή τη δευτερογενή μετανάστευση. Η Τσεχία, για παράδειγμα, είχε ε, μερικές δωδεκάδες ε, που πήγαν στη χώρα που μέσα σε ένα μήνα φύγανε και φύγανε για τη Γερμανία. Εμείς τους συμπεριφερθήκαμε υπέροχα. Και πρέπει να σα πω πω αφήσαμε και τα παιδιά του να πάνε σχολείο και φύγανε για τη Γερμανία. Τέταρτη ερώτηση. Διάβασα τη σύμβαση τη Γενέβη. Και αυτό μάλλον με κάνει διαφορετικό από του υπόλοιπου. Το να μεταφέρονται τα άτομα αυτά ε, μέσα στην Ευρώπη δεν ε, έρχεται σε αντίθεση με τη σύμβαση της Γενέβης. Εγώ δεν έχω το κείμενο μπροστά μου, αλλά λέει, αν θυμάμαι καλά, πως κανένα άτομο δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να ζει σε συγκεκριμένη χώρα. Πέμπτη ερώτηση. Όταν θα λάβει χώρα αυτή η δευτερογενής ε, μετανάστευση, ποιος θα είναι υπεύθυνο. Οι Γερμανοί δεν ξέρουν αν τα άτομα αυτά που μετεγκαταστάθηκαν στην Τσεχία θα φτάσουν σε αυτούς, θα τους στείλουν πίσω στην Τσεχία ή θα τους στείλουν πίσω στο Ιράκ. Είναι μια γελία νομική κατάσταση. Ερώτηση 6. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε το τράφικινγκ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίζει ποιος θα μεταφερθεί και πού. Γιατί στην κομμουνιστική εποχή στην Τσεχία λέγαμε έναν έκδοτο και λέγαμε αν λέω ψέματα, να με πάρει ο αέρας και να με πετάξει στη Δυτική Γερμανία ε, για να τιμωρηθώ. Και βέβαια όλοι λέγανε ψέματα για να καταφέρουν να φτάσουν στη Δυτική Γερμανία. Ε, τι θα γίνει αυτό με τα hot spots στην Ελλάδα. Όλοι θα θέλουν να πάνε στη Δυτική Γερμανία ή στη Σουηδία. Κανείς δεν θα θέλει να πάει στην Τσεχία. Και έχω μιλήσει με πολύ κόσμο. Και η έβδομη ερώτηση είναι η εξή. Και πρέπει να σα πω, σε... καταλαβαίνω και εκτιμώ αυτά που κάνετε. Και καταλαβαίνω τα όσα κάνει και η κυρία Γιώτοβα που πήγε και αποστολή στη Σικηλία. Οπότε η φιλοσοφική ερώτηση που έχω να σας θέσω τώρα είναι και δεν χρειάζεται να απαντήσετε αμέσω. είναι η Ιαπωνία δέχθηκε 15 πρόσφυγες πέρσι. Δείχνει αλληλεγγύη η Ιαπωνία με την Ευρώπη, με τους πρόσφυγες ή είναι ξενόφοβοι. Μαντάμ Ουίσμπερκ. Η ειναι ξενοφοβοι Ουίσμπερκ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Θα χρειαστεί χρόνος, ναι. Από ό,τι ακούμε γύρω στα τρία χρόνια θα αναθεωρηθεί ε, το ε, Δουβλίνο, ε, η συνοριοφυλακή, ε, το ΕΚΑΣ, όλα αυτά ε, που χρειάζονται να γίνουν. Αλλά από ό,τι βλέπω στη χώρα μου η κατάσταση είναι χαοτική, γιατί εμείς υποδεχόμαστε πάρα πολύ κόσμο. Έχω λοιπόν μια ερώτηση για το Δουβλίνο 3 και για τους ανθρώπους που έρχονται μόνοι. Θα πρέπει να τους ρωτάμε πού πρέπει να πάνε. Ε, φυσικά ε, μπορεί να μην ε, γίνει δεκτό το αίτημά τους, αλλά θα πρέπει να τους ρωτάμε. Στην Σουηδία έχουμε, έχουμε υποδεχτεί 35.000 νέους άντρες πέρυσι, ασυνόδευτους πρόσφυγες. Πώς θα τους διανύμουμε μεταξύ των κρατών μελών, τι θα κάνουμε ε, κάποιες ε, εξετάσεις, ε, να δούμε πόσο ετών είναι, για παράδειγμα, για να τους πάμε δεξιά και αριστερά. Αν θέλουμε να τους στείλουμε, ας πούμε, στην Τσεχία, ίσως ε, να μην ε, είναι το καλύτερο μέρος για αυτούς και να θέλουν να πάνε στη Σουηδία. Υπάρχει ένας συνάδελφος από την Τσεχία που ανέφερε και το κόστος της μεταφοράς ε, ε, για αυτούς τους ανθρώπους. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν είναι έτοιμα για μια κοινή πολιτική ασύλου και γι' αυτό δεν συμβαίνει τίποτα, δεν βλέπουμε καμία πρόοδο. Πολλά κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα γιατί δεν το θέλουν. Πρέπει να το δούμε λοιπόν αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Όνσπερκ. Ο κύριος Αλάχο έχει τώρα το λόγο. Thank you, Madam Chair. Αλάχο, λοιπόν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι διάφορες ε, εθνικότητες έχουν διαφορετικό βαθμό αναγνώρισης στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η δευτερογενής, ας πούμε, κίνηση, η επιλογή ασύλου ε, έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία πέρασαν από την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Γερμανία και την Δανία για να ζητήσουν άσυλο στην Σουηδία και στην Φιλανδία. Οι πιθανότητες ενός ετούντος άσυλο να αναγνωριστεί ε, ως πρόσφυγας εξαρτάται από τη χώρα που είναι υπεύθυνη να επεξεργαστεί το αίτημά του. Το πρόβλημα αυτό θα παραμείνει. Ακόμα και όταν αναθεωρηθεί το σύστημα του Δουβλίνου. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο κίνητρο για έναν παράνομο μετανάστη να μην ε, καταγραφεί στην πρώτη χώρα εισόδου. Χωρίς τους εσωτερικούς ε, συνοριακούς ελέγχους δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά ε, για τους ανθρώπους που μπορούν άμεσα να περάσουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο για να καταθέσουν αίτηση ασύλου ή να πάνε σε ένα άλλο ε, κράτος όταν έχουν ήδη πάρει άσυλο. Οι άνθρωποι φτάνουν στην Ιταλία και στην Ελλάδα όχι γιατί θέλουν να μείνουν εκεί, αλλά γιατί ξέρουν ότι από εκεί μπορούν να περάσουν στο βορρά. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν έχει νόημα να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη αυτόματα να απορρίπτουν αιτήματα από άτομα που έρχονται ξεκάθαρα από άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα μειώσει και την πίεση στην Ελλάδα και την Ιταλία κατά τη γνώμη μου. Γιατί ε, οι χώρες αυτές για τους περισσότερους μετανάστες είναι χώρες διέλευσης. Ευχαριστώ τον κύριο Λάχο. Ο κύριος Ράντεφ είναι ο τελευταίος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μισελ για την παρουσίασή σας. Ε, να πω ότι αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απάντηση απλώς ε, στα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το έγγραφό σας, οι ετούντες άσυλο θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην πρώτη χώρα που καταφτάνουν και κατά αυτόν τον τρόπο η χώρα αυτή θα είναι υπεύθυνη για αυτούς. Αυτό δεν θα αλλάξει την κατάσταση που ισχύει τώρα ε, για την Ελλάδα και για τη Βουλγαρία, ας πούμε, ε, στο μέλλον ενδεχομένως. Η τρέχουσα κρίση έχει δείξει ότι το σύστημα δεν λειτουργεί και πρέπει να αλλάξει. Είναι ξεκάθαρο ότι τα άτομα αυτά δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα που φτάνουν. Θέλουν να πάνε στη Γερμανία ή γενικά στις σκανδιναβικές χώρες. Δεν έχετε λοιπόν προτείνει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει βέβαια αυτή η αλλαγή στην έννοια της οικογένειας. Προσθέσατε τα αδέρφια και τους συζύγους ε, ε, όταν ε, ο γάμος έχει συνηθεί μετά την άφηξη. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακαλύψουμε ότι όλες αυτές οι αφήξεις έχουν κάποιο συγγενή. Και έχουν κάποιο λόγο να ε, έχουν την διεθνή προστασία. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν και κάποιοι γάμοι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Κάτι άλλο. Αυτοί που δεν έχουν έγγραφα για να αποδείξουν την ταυτότητά του, ε, κατανοείται ε, ότι οι γάμοι που γίνονται στα ε, στρατόπεδα των προσφύγων ε, δεν γίνονται βάση πιστοποιητικών και ούτε ενώπιον επίσημων αξιωματούχων. Δεν θα δεστρεβλώσει αυτό το σύστημα. Ευχαριστούμε κύριε Ράντεφ και τώρα μετά τις ερωτήσεις που τέθηκαν θα μπορούσατε να μας δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις για το κατά πόσον πρόκειται για μια ριζοσπαστική πραγματικά μεταρρύθμιση όπως είχαμε ακούσει τόσες φορές εδώ και καιρό και τη ζητούσαμε. Αυτά που μας προτείνατε βάσει των συναδέλφων και των απόψεών τους είναι καλοπιστικές αλλαγές ε, ο μηχανισμός που προτείνατε δεν θα δουλέψει. Δεν θα δουλέψει όπως είχε συμβεί και στην προηγούμενη περίπτωση, με το προηγούμενο σύστημα. Τι γνώμη έχετε λοιπόν γι' αυτό. Ε, πώς θα λειτουργεί αυτός αυτόματος, αυτός αυτόματος μηχανισμός που απολογεί τον αριθμό των ε, ατόμων. Ε, μιλάμε για ζωντανά άτομα, για ανθρώπους, για ένδια το θέμα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να περάσουν τα σύνορα και δεν μπορούν να τους καταγράψουν καν οι σύνοριοφύλακες. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Αν ακούσετε τις απόψεις των διαφόρων ε, συναδέλφων, Υπάρχουν πολλά αντιφατικά σχόλια. Γιατί δεν είναι απλό ακριβώς. Όντως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, με ανθρώπινα όντα. Θέλουν να μετακινηθούν, να πάνε στη Γερμανία, στη Σουηδία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν πάρουμε τη δεύτερη επιλογή σε σχέση με τις προτάσεις και πάλι θα έχουμε δεύτερο γενείς μετακινήσεις. Ό,τι επιλογή και να προκρίνουμε, θα έχουμε δευτερογενεί μετακινήσει. Επιλογή 2, 3, 4, όποια εφάνταστη λύση και να βρείτε, οι άνθρωποι θα θέλουν να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα σύστημα το να είναι δίκαιο για τα κράτη-μέλη και το οποίο να καταστά σαφέ και στου μετανάστε ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν και τελείω ελεύθερα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει σύγκληση στα συστήματα ασύλου μα. Θα συμφωνήσω με την κυρία Βίξτρεμ. Πρέπει να το βλέπουμε σφαιρικά το θέμα και να βεβαιωθούμε ότι το πακέτο θα παρουσιάσει συνεκτικέ νομοθετικέ προτάσει. Ε, όλα τα νομικά κείμενα να προχωρήσουν παράλληλα, να συμβαδίσουν. Ο κόσμο θα συνεχίσει να μετακινείται δευτερογενώ. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τι δευτερογενεί μετακινήσει. Πρέπει να το δεχτούμε. Όμω, αν περιορίσουμε το δικαίωμα των ανθρώπων που δεν εφαρμόζουν του κανόνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον θα λειτουργήσει αυτό αποτρεπτικά. Πρέπει να εξηγήσουμε στους μετανάστες ότι υποτίθεται ότι δραπετεύετε για τη ζωή σας. Σας προστατεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορείτε να διαλέγετε και το κράτος μέλος. Εάν θέλετε και να διαλέξετε, θα σας στείλουμε πίσω. Και θα χάσετε κάποια δικαιώματα ως προς τα ημερήσια επιδόματα και το καθεξής. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν παραβιάζουν το σύστημά μα. Ιδάλω ποτέ δεν θα υπάρξει ένα ευρωπαϊκό, κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Αυτό που προτείνουμε δεν είναι καλοπιστικέ αλλαγέ. Είναι επί τη ουσία αλλαγέ. Διότι δημιουργούμε de facto ένα μόνιμο σύστημα επανακατάστασης. Το 150% σαν το όριο θα, ε, είναι ένα όριο που θα φτάσουν πολύ γρήγορα στην Ελλάδα. Δείτε τους αριθμούς, το, ανα, το ΑΕΠ, τον αριθμό των κατοίκων και το πώς οι μετανάστες φτάνουν. Ακόμη και τώρα, σήμερα να το εφαρμόζαμε, θα φτάναμε το όριο, ακόμα και με τις περιορισμένες αφήξεις. Αλλά αν υπάρχει ένα διαρκές σύστημα επανεγκατάστασης για την Ελλάδα, δεν απέχουμε και πάρα πολύ από την επιλογή 2. Η επιλογή 2 όμως δεν πρόκειται να περάσει στο Συμβούλιο. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε κάπως επικοδομητικοί εδώ ε, με το Συμβούλιο. Έχουμε αυτά που ζητάτε. Τα ζητάτε εδώ και χρόνια στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Το λέτε, ναι, ένα δίκαιο σύστημα με αλληλεγγύη. Ο μόνος τρόπος όμως να γίνει είναι να φτάσουμε σε συμβιβασμό στο Συμβούλιο. Το γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο είναι και αυτό διχασμένο. Πρέπει λοιπόν να πετύχουμε ενότητα και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για να φτάσουμε σε μια λογική συμβαστική λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε όλε τι θέσει. Πιστεύει ότι αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο. Η επιλογή ένα είναι ο καλύτερο τρόπο να φτάσουμε το στόχο μα. Πρέπει να κοιτάζουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα, στην πράξη. Εκεί να δούμε αν μπορούμε να αποτρέψουμε τι δευτερογενεί μετακινήσει. Και συμφωνούμε με την κυρία Βίξτρομ. Χρειάζεται κάτι που να είναι λειτουργικό. Ευχαρίστω λοιπόν να εργαστούμε σε τεχνικό επίπεδο, να εξηγήσουμε πώ θα λειτουργεί το σύστημα, να εξηγούμε ποιο θα πληρώνει το κόστο των μετακινήσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασιστεί αν θα καλύπτει το κόστος των μετακινήσεων, το κόστος της επανακατάσταση, Για όσου ε, μετακινούνται δευτερογενώ θα είναι ευθύνη των κρατών μελών στο σημείο άφηξης δηλαδή, να τους στέλνουν πίσω εκεί που θα έπρεπε να αποσταλούν. Αυτό συμβαίνει και τώρα βάσει του Δουβλίνου. Οι άνθρωποι αποστέλλονται πίσω και το κόστο το καλύπτει το αρμόδιο κράτο μέλο. Μπορούμε να το σκεφτούμε κι άλλο, να βρούμε κατάλληλε λύσει. Εδώ είμαστε ευέλικτοι, αλλά πρέπει να υπάρχει αυτό ο διαφορετικό μηχανισμό. Εάν περάσει στο Συμβούλιο, θα είναι μείζον νίκη και επίτευγμα για το σύστημά μας. Για τις προτιμήσεις των ετούντων άσυλο. Εντάξει, το σκεφτήκαμε πολύ. Δεν ε, τους αρνηθήκαμε ομά κάθε δικαίωμα, τα σκεφτήκαμε πολύ προσεκτικά. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Με γλωσσικές δεξιότητες. Έχουμε τούντες άσυλο που λένε ότι Θέλω να πάω στην Πολωνία γιατί μιλάω πολωνικά. Φτάνοντα στην Ελλάδα. Πώ θα το ελέγξει κανεί αυτό. Μαθήματα, δάσκαλοι. Πού να του βρούμε. Και ποιο θα είναι το επίπεδο επάρκεια στα πολωνικά για να πει κανεί αυτό ο άνθρωπο μπορεί να πάει στην Πολωνία. και όχι στη Δημοκρατία τη Τσεχία. Για σκεφτείτε λιγάκι πόσε λεπτομέρειε έχει ένα τέτοιο σύστημα τι επίπεδο πολωνική γλώσσα θα απαιτείται για να πάει ένα άνθρωπο ε, στην Πολωνία. Προσόντα, επαγγελματικά προσόντα. Πώ θα τα αντικαταστοιχίσουμε με τι απαιτήσει των κατομελών, πώ θα κοιτάξουμε τα πτυχία. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα επαναγκατάσταση που να λειτουργεί. Είδαμε του τελευταίου μήνε ότι είδο, ήδη, όταν θέλουμε να επαναγκαταστήσουμε του ανθρώπου, έχουμε πάρα πολύ μεγάλε δυσκολίε. Μην το κάνουμε πιο περίπλοκο. Α το κάνουμε λίγο απλό, ευέλικτο και ταχύ στην εφαρμογή του. Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει δραστικά το σύστημα. Τέθηκαν κάποιε φιλοσοφικέ ερωτήσει για την Ιαπωνία. Θα συμφωνήσω απολύτω με όσα είπατε. Η Ιαπωνία πρέπει να πάρει περισσότερου. Θα πρέπει να εμπλακεί στην επαναγκατάσταση. Νομίζω ότι η διάσκεψη που κάλεσε ο πρόεδρος Ομπάμα στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο επίσης μπορεί να φέρει περισσότερες υποσχέσεις και από άλλες χώρες, οι χώρες του κόλπου, η Ιαπωνία ίσως, να πάρουν και αυτοί κάποιους ήρους. Είναι πολλοί οι, διεθνεί εταίροι, οι διεθνείς εταίροι που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα. Για τον έλεγχο των εσωτερικών συνόρων. Δεν νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε τον ε, έλεγχο των ιστορικών σύνορων. Διότι με το σύστημα των hot spot, όπω περιγράφει προηγουμένω, ο καθένα θα καταγράφεται. Θα έχουμε κόσμο που θα είναι καταγεγραμμένο στην πρώτη χώρα, τη χώρα τη πρώτη αύξηση, και μετά θα είναι καταγεγραμμένο καταχωρισμένο στο σύστημα. Εάν υπάρξει δευτερογενή μετακίνηση, θα εμφανίζεται αυτό στο σύστημα. Και η χώρα στην οποία θα αποστέλλεται επίση θα εμφανίζεται στο σύστημα. Οπότε θα είναι αρμοδιότητα του εν λόγω κράτου μέλου να ασχοληθεί με την απερικατάσταση. Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει το VIS, το VIS. Ε, είναι ένα σύστημα απλό, εύχριστο και λειτουργικό. Έτσι το έχουμε σχεδιάσει. Βεβαίω να το τροποποιήσουμε εφόσον χρειαστεί. Εάν ε, καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα μα στι συζητήσει με το Ευρωκοινοβούλιο, είμαστε ανοιχτοί σε ιδέε, σε βελτιώσει, αλλά συζητούμε με τον κόσμο και οι άνθρωποι θέλουν να φτάσουν σε μια χώρα προορισμό, αλλά εάν του ρωτήσει κανεί με λεπτομέρειε, γιατί θε να πα στη Γερμανία, δεν ξέρουν. Δεν έχουν απάντηση. Πραγματικά δεν έχουν απάντηση. Απλώ του το έχουν πει οι διακινητέ, έτσι του έχει έρθει ιδέα. Ε, νομίζω ότι έτσι θα βρουν δουλειά. Όταν καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλάζει η γνώμη του. Εάν δείτε τώρα, υπάρχουν πολλοί Αφγανοί και Ιρακινοί που ζητούν εθελοντικά να επιστρέψουν. Συνειδητοποιούν αυτό που του υποσχέθηκαν οι διακινητέ δεν ήταν πραγματικό. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να ε, έχουμε και συμμετοχή των ίδιων των μεταναστών, να τους πείθουμε. Αυτό κάνουμε τώρα με το σύστημα της επανακατάστασης. Ε, βλέπουμε όλο και περισσότεροι να είναι πρόθυμοι να επανακατασταθούν. Δεν είναι λοιπόν ένα σύστημα μόνο μαθηματικό ε, στεγνό το οποίο απλώς θα εφαρμοστεί. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να υπάρξει διαρκής ε, παροχή στήριξη στους μετανάστες Καθόλου τη διάρκεια της διαδικασίας να τους ενημερώνουμε όταν φτάνουν, όταν έρχονται και μετά συστηματικά για το πώ λειτουργεί το σύστημα. Δεν αντίκειται στη σύμβαση τη Γενέβη το σύστημα. Ίσα ίσα. Η σύμβαση τη Γενέβη μιλάει για την αρχή τη μία επαναπροώθηση προ μία χώρα που δεν είναι ασφαλή. Εδώ μιλάμε για επανακατάσταση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρε που υποτίθεται είναι εντό των κριτηριών τη σύμβαση τη Γενέβη. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανεί δεν μα επικρίνει γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μουσόλ. Ε, θα κάνω μια εξαίρεση για την κυρία Μετσόλα, η οποία είναι συγκέντρια και μόλις έφτασε. Ε, και υπάρχουν και εκθέσεις και πάλι σε επιτροπές. Κυρία Μετσόλα, για δύο λεπτά σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βίκστρομ και να πω σε σχέση με τα πόσα ακούστηκαν προηγουμένως ότι θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση για να δούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε με αυτό το φάκελο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι η δική μου χώρα που αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και η αντιμετώπιση που έχουμε από την πλευρά του ΕΛΚ αποδεικνύει πως το σύστημα του Δουβλίνου δεν λειτουργεί. Και τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης αντιμετωπίζουν τεράστιες πιέσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ολόκληρη αναθεώρηση του συστήματος, μια σφαιρική αναθεώρηση ε, για να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει το κοινοτικό κεκτημένο. Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και όπου θα συνεργαστούμε και με την εισηγήτρια και με την Κομισιόν για να βρούμε μια λύση η οποία ενδεχομένως να μπορεί να ε, γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Και κλείνοντας να σας πω πως ε, θέλουμε να κάνουμε όσο μπορούμε, όσο μπορούμε για να αποθαρρύνουμε αυτή τη δευτερογενή μετακίνηση όπως είπατε και εσείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Madame Metzola, Madame est est-ce Ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Μιλήσατε πολύ και με λεπτομέρειες. Θέλετε όμως παρόλα αυτά να ξανααπαντήσετε. Έχετε άλλες, άλλα σχόλια να κάνετε. Ε, ευχαριστώ. Τα πιο σημαντικά τα είπα. Αλλά θα ήθελα να στραφώ εκ νέου στους συναδέλφους, μια που ήρθε και η Ρομπέρτα στην αίθουσα, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μείνουμε μια ομάδα ενωμένη και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα προς ένα συμπληκτικό και ανθεκτικό σύστημα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα συνεχίσουμε το διάλογο που γίνεται μεταξύ μας για να βρούμε μια κοινή θέση. Βήμα-βήμα, επαναλαμβάνω, όταν δούμε και τους άλλους φακέλους πώς προχωράνε και να ε, στραφούμε προς τα κράτη-μέλη που είναι μακριά από τη δική μας θέση στο Ευρωκοινοβούλιο και να τους πούμε ότι κοιτάξτε δεν έχει για το αν θα κάνουμε ε, κάτι το οποίο θα κλείσει ε, θετικά. Είμαστε υποχρεωμένοι. Στη ζωή καμιά φορά υποχρεούσα να κάνεις κάποια βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και ε, εύχομαι να συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Μουσέλ. Euh, alors, το επόμενο σημείο είναι και το τελευταίο της ημερήσιας διάταξης. Φτάσαμε στην παρουσίαση της εισηγήτριας της κυρίας Μαγιον, Φαγιών του σχεδίου έκθεσης κατάλογος τέτος χωρών ε, για ε, την ε, εξαίρεση του κοσυφοπεδίου από τον κατάλογο των τρίτων χωρών, των οποίων, στον οποίο οι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρηση, αρκεί να υπάρχουν ε, βιομετρικά διαβατήρια. Αυτό πέρασε από την Επιτροπή μα τον Μάιο και το συζητήσαμε και με εκπροσώπου του Κωσυφοπεδίου βάσει μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012. Ο διάλογο για τι θεωρήσει ε, διεξήθη χωρί να επηρεάσει τι απόψει των κρατομελών για το καθεστώ αναγνώριση του Κωσόβου. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα την παρουσίαση της για ε, έκθεση από την εισηγήτρια και μετά θα ακούσουμε και τους σκιώδεις εισηγητές. Ο λόγος στην κυρία Φαγιών. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση για το κοσυφοπέδιο είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα, διότι είναι μια νεαρή κοινωνία η οποία μας κοιτά με τα μάτια γεμάτα ελπίδα. Νομίζω ότι όλοι αυτό το γνωρίζουμε. Ξέρω πολύ καλά τη χώρα, ξέρω την περιπλοκότητα και την ευαισθησία της. Ε, είμαι ιδιαίτερα περήφανη που μπορώ να παρουσιάσω μια έκθεση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων λόγω της πρόοδου που έχει πετύχει η χώρα τελευταία. Μερικοί μπορεί να λένε γιατί βιαζόμαστε. Γιατί η απάντησή μου είναι ότι αυτή η χώρα έχει παραμείνει απομονωμένη για πάρα πολύ καιρό υπέρ το δέον και έχει ε, εκπληρώσει πάνω από 90 όρους ε, για να μπορεί να έχει αυτή την απελευθέρωση, πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Σήμερα οι πολίτες μπορούν να πάνε χωρίς βίσα μόνο σε τέσσερις ευρωπαϊκές αυτό είναι μια απομόνωση που επηρεάζει την καθημερινή ζωή των πολιτών, ειδικότερα των νέων, γιατί αυτού έχω πρώτα στο μυαλό μου όταν μιλάω για την κατάργηση των θεωρήσεων. Θέλω να του δώσω την ίδια ευρωπαϊκή προοπτική που οι νέοι στην ε, περιφέρεια αυτή που καταστράφηκε από του αιματηρούς πολέμους ήδη απολαμβάνουν. Ε, όσο περισσότερο κρατούμε λοιπόν αυτή τη χώρα στην απομόνωση, τόσο περισσότερο δίνουμε πρόσφορο έδαφος στο οργανωμένο έγκλημα που ε, δίνει παράνομα έγγραφα. Για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής ε, πρέπει να προχωρήσουμε στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της άμεσης γειτονιάς της. Είναι ε, θέμα η αναγνώριση από τα πέντε κράτη-μέλη και ελπίζω σύντομα να δούμε πρόοδο, αλλά αυτό δεν αποτελεί ώρα για την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ξεκάθαρη. Το κοσυφοπαίδιο πληρεί τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση, τον αδικό χάρτη δηλαδή, και τα δύο στοιχεία που απομένουν να γίνουν θα έχουν ε, εφαρμοστεί πριν την έγκριση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να αναφέρω το πιο σημαντικό. Είναι επίγον το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου να κυρώσει τη συμφωνία ε, με, για την ε, ε, καταγραφή των συνόρων με το Μαυροβούνιο. Αυτό έχει γίνει ένας νέος όρος που προέκυψε κατά την διαδικασία και έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα το κάνει. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε την απελευθέρωση όπως είπα. Το Κωσυφοπαίδιο έχει θεσπίσει ένα σύγχρονο και λεπτομερές σύστημα για την ανείχνευση των εγκληματικών διαδικασιών που ήδη έχει αποφέρει καρπούς. Επίσης είμαι πεπισμένη ότι οι νέες τεχνολογικές πράξεις όπως τα βιομετρικά διαβατήρια που απαιτούνται θα μας δώσουν μια δυνατότητα να έχουμε πιο ακριβείς ελέγχους στα σύνορα. Η ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους σχετικούς οργανισμούς θα μας βοηθήσει να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών για πιθανές απειλές. Να καταλήξω θυμίζοντας σε όλους ότι η απελευθέρωση από τις θεωρήσεις αποτελεί ένα απτό βήμα για τους πολίτες μας, ειδικά για τους απλούς πολίτες και τους νέους ανθρώπους οι υπόλοιποι, ε, για να είμαι ειλικρινή, θα βρουν τρόπο να ταξιδέψουν. Είναι επίση σημαντικό η απελευθέρωση των θεωρήσεων να έχει κάποιου περιορισμού, να το γνωρίζει ο κόσμο. Και κάθε φορά που ε, ταξιδεύω και πηγαίνω στο 25, αυτό το αναφέρω. Ενισχύουμε τον ε, μηχανισμό για προσωρινή αναστολή του μηχανισμού θεωρήσεων αυτές τις εβδομάδες και θα μπορεί κανείς να αντιδράσει σε περίπτωση παραβιάσεων. Στην περίπτωση λοιπόν της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιούμε πότε υπάρχει πρόοδος, πότε πληρούνται κριτήρια από χώρε και να ενισχύουμε τις προσπάθειες να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ μόν και των άλλων πολιτών. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η συνεργασία με το κοσυφοπαίδιο, οι κοινέ προσπάθειες να φέρουμε το κοσυφοπαίδιο πιο κοντά σε εμάς ε, και η προσπάθεια να κλείσουν τα εκκρεμή ζητήματα θα ε, στεφθεί με επιτυχία πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φαγιών και τώρα λόγω στου κοιόδης εισηγητές από το ΕΛ και κυρία Κάμπριελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ευχαριστούμε την κυρία Φαγιών για την παρουσίαση του σχεδίου έκθεση. Όλοι συμφωνούμε Υπάρχουν σοβαρέ ιδέε που διατρέχουν όλο το κείμενο και ναι, πρέπει να θυμίσουμε όταν μιλάμε για απελευθέρωση καθεστώτο θεωρήσεων να απευθυνόμαστε στου πολίτε. Χρειάζεται να προβάλλεται η εταιρική μα σχέση με το κοσφό πεδίο για να περάσει και ένα μήνυμα προ του πολίτε το οποίο είναι σαφέ. Ναι, θέλουμε απελευθέρωση του καθεστώτο των θεωρήσεων, όμω από την άλλη είναι σαφέ ότι η αξιοπιστία μα ω Ευρωκοινοβουλίου ε, συνδέεται άμεσα με το σεβασμό όλων των κριτηρίων. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο θέλω να επιμείνω στο εξής Υπάρχει ανάγκη να γίνονται πλήρως σεβαστά τα δύο εναπομείναντα κριτήρια. Είναι ε, σοβαρό για μας όταν επιμένουμε στα δύο αυτά κριτήρια να επιμένουμε ταυτόχρονα και στην εξής ιδέα. Ως κοινοβούλιο δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε ασυνέπειες που μπορεί να παρερμηνευθούν κατά την υλοποίηση των αρχών του πλήρου σεβασμού των κριτηρίων. Ε, εξαρτάται από αυτό η αξιοπιστία μας, αλλά και η, αξιοπιστία των προσπαθειών του κοσφοπεδίου και των χωρών που είναι στην ε, οδό, στην άγουσα ε, ή κοντά στο στόχο της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Πρέπει λοιπόν να δούμε σημαντικά βήματα πρόοδου ε, πριν προχωρήσουμε τη διαδικασία. Ναι, για τη διαχείριση των σύνορων, ναι, ε, στο τι έχει γίνει στα σύνορα με το Μαυροβούνιο, αλλά υπάρχει και μια απόφαση τη 15 η Μαρτίου, ε, σύσταση διεθνου επιτροπη και αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση της είναι πολύ σημαντική και να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια από τι αρχέ που είναι ένα από τα θεμέλια ε, των ιδεών, των αρχών που μας ενώνουν, είναι ότι δεν θα έχουμε καμία ε, αμφισβήτηση, καμιά εδαφική ακεραιότητας, κανενός τους μέλους. Και δεύτερον, καταπολέμηση του εργανομένου εγκλήματος. Εκτιμούμε τι προσπάθειε που γίνονται προ αυτή την κατεύθυνση, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να έχουμε αποτελέσματα διαρκεία, βιώσιμα. Είναι και αυτό μια προπόθεση για την απελευθέρωση του καθεστώτο θεωρήσεων. Υπ' αυτήν την έννοια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω να μπορεί να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε σε ό,τι αφορά τι βασικέ αυτέ δυσκολίε που πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού να πούμε σαφώ ότι εντάξει, τα κριτήρια αυτά πληρούνται. Και Τέλος, έχω επιμείνει πολύ στα κριτήρια αυτά, ακριβώς γιατί δεν κρύβουμε τον προβληματισμό μα για την αναγνώριση του νομικού καθεστώτο του κοσυφοπεδίου από τα κράτη-μέλη. Να πω ότι ακόμη πέντε κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν ε, το κοσυφοπέδιο ω ανεξάρτητο κράτο και πρέπει να παραμένουμε πολύ συνετοί ε, και να είμαστε προσεκτικοί. Όταν μιλάμε για καθεστώ, μιλάμε και για έγγραφα ταυτοποίηση, τα οποία ε, συνδέονται άμεσα με τα ταξίδια που επιχειρούν να κάνουν οι πολίτε Πάντω, παρόλα αυτά, αναφέρεται στην εκθεσή σα και συγχαρητήρια κυρία Φαγιών ότι πέντε τη μέλη ασχολήθηκαν με τη διαδικασία απελευθέρωση του καθεστώτο θεωρήσεων για το κοσμοπέδιο υπό την αίρεση συμπλήρωση των, ε, πλήρωση μάλλον των κριτηρίων, χωρί όμω αυτό να επηρεάζει το καθεστώ αναγνώριση του κοσμοπαιδίου. Ναι, επιμένω κι άλλη μια φορά ότι τα κριτήρια πρέπει να πληρούνται πλήρω. Είναι λοιπόν καθήκον μα πολιτικό με το εργαλείο τη απελευθέρωση των θεωρήσεων να ενισχύσουμε την εταιρική μα σχέση με το κοσμοπέδιο προ όφελο των πολιτών, όμως, εξίσου ευθύνη μας είναι να παραμείνουμε αξιόπιστοι, σεβόμενοι την αρχή ε, συμπλήρωσης όλων των κριτηρίων με πρώτερη προϋπόθεση την κλήψη ε, ε, υπόψη των αποκρουσών που είναι τόσο σημαντικές για μας. Ευχαριστώ. Οι διερμηνείς είναι πολύ ευγενείς, μας έδωσαν λίγα λεπτά παραπάνω, αλλά σας παρακαλώ δύο λεπτά ανά άτομο. κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο εξ ονόματος της συναδέλφου Μαρή Κριστίν Βερζιά, ε, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Για την ομάδα μας. Βεβαίω και είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων. Είναι σημαντικό. Όμως επιμένουμε ότι όλα τα κριτήρια πρέπει να γίνουν σεβαστά. Είναι 98 στην περίπτωση του κοσφοπεδίου και αφορούν θέματα που ήδη αναφέρθηκαν. Διαφθορά, οργανωμένο έγκλημα, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλος ιδιαίτερα στον Ρωμά. Ε, Για αυτόν το λόγο Καλώς υπενθυμίστηκε σε αυτό το πλαίσιο ότι υπάρχει ψηλό ποσοστό ε, πολιτών του κοσμοπεδίου, οι οποίοι έχουν λάβει ε, διεθνή προστασία σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στη Γαλλία. Άρα υπάρχουν κριτήρια τα οποία δεν γίνονται ακόμη σεβαστά. Στις 7 Μαρτίου το 2016, η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης θύμισε ότι το πεδίο χρειάζεται ακόμη ανεξάρτητους μηχανισμούς για να ελέγχει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη και τώρα τελευταίος ο, ο κύριος Μπούχνερ, αν σωστά προφέρω το όνομα. Thank you, uh, Ευχαριστώ πολύ. Εδώ εκφράζομαι εκ μέρους της κυρίας Λούνατσεκ, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί σήμερα, διαβάζω το κείμενό της. Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την πολύ αναμενόμενη απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συστήσουμε μια απελευθέρωση υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες του κοσμοπεδίου. Τονίζουμε την μεγάλη σημασία της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για τους πολίτες του κοσμοπεδίου. Επιθυμούμε να έχουμε μια σύντομη κατάληξη της διαδικασίας και θέση σε εφαρμογή του τροποποιημένου κανονισμού το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να διευκολυθούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον, ειση... τον εισηγητή που αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της πρότασης και για το πολύ ε, ε, φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο έκθεσης. Για να μην καθυστερήσουμε παραπάνω την ε, διαδικασία δεν θα υποβάλουμε καθόλου τροπολογίες. Η απελευθέρωση από την υποχρέωση θεώρηση είναι ο τρόπος που θα προωθήσει τις επαφές μεταξύ ανθρώπων και θα διευκολύνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε μια εποχή όπου η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται. Το Κωσυφοπέδιο είναι η μόνη χώρα από τα Βαλκάνια που από το 2010 εξακολουθούν να μην μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρώπη παρόλο που από το 2010 ελευθερώθηκε το ταξίδι για, όλο τους, για όλους τους υπόλοιπους πολίτες των Βαλκανίων και χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο που έχει δημιουργήσει την εντύπωση στον πληθυσμό πως είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και πως είναι κλειδωμένοι στη χώρα τους. Εμείς καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να εφαρμόσουν γρήγορα τις ε, εναπομείνουσες δύο προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση να παρουσιάσει ε, όλο τον κατάλογο των καταδικών που χρειάζεται για τα θέματα διαφοράς, διαφθοράς και ε, Ε, οργανωμένου εγκλήματος και δεύτερον για την ε, η αντιπολίτευση και τη Βουλή να υπογράψουν την επικύρωση της χάραξης των γραμμής των συνόρων ε, και της μεθορίου με το Μαυροβούνιο. Θα πρέπει λοιπόν το Κωσυφοπέδιο να λάβει αυτή την χωρί, την απελευθέρωση. Κύριε Πίχνερ, δεν έχετε άλλο χρόνο. Θα δώσω τώρα το ρόλο, το λόγο στην κυρία Σμιτ που ε, εκπροσωπεί εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, thank you very much. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γρήγορη προετοιμασία της ε, ε, έκθεσης και την υποστήριξη της πρότασης της Επιτροπής. Εμείς ε, ε, υποστηρίζουμε την πρόθεση της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην πλήρωση των δύο εναπομείναντων ε, κριτηρίων για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, η οποία θα γίνει μόλις πληρωθούν όλα τα κριτήρια. Ο συνάδελφος Μπενεντέκο από τη Γενική Διεύθυνση HOME θα σας ενημερώσει στα γρήγορα για το τι συμβαίνει σχετικά με αυτά τα δύο κριτήρια που απομένουν. Ευχαριστώ, Γκάβη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω λίγα λόγια για τα δύο στοιχεία που απομένουν να γίνουν, όπως αναφέρθηκαν. Ξέρουμε από την κυβέρνηση ότι υπάρχει πλήρης δέσμευση για κύρωση των συμφωνιών με το Μαυροβούνιο αν είδατε τις ειδήσει, ε, εσωτερικά το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή και να, μιλήσουμε, να μιλήσουν οι διάφοροι πολιτικοί ε, μεταξύ τους, έτσι ώστε όταν κατατεθεί το σχέδιο κύρωσης να διασφαλιστεί η κύρωση. Άρα ο χρονισμό είναι στα χέρια της κυβέρνησης, αλλά η κυβέρνηση έχει αναλάβει πληρώ τη δέσμευση κύρωση τη συμφωνία, η οποία βασίζεται σε μια μακροχρόνια διαδικασία ε, των συνόρων με το Μαυροβούνιο. Τώρα, ε, για να δούμε ε, στο παρελθόν, ε, το ε, μπορούσε να ανοιχνεύσει πολλές περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος 30 30%, ε, 30 ε, ε, περίπου περιπτώσεις, τώρα έχουμε φτάσει στο 35 το νούμερο. 17 ήταν η, οι διώξεις και υπάρχει η απαγγελία κατηγοριών συγκεκριμένα και σε αυτές τις περιπτώσεις ε, ε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αποτελέσματα. Αν δούμε ακριβώς ε, τι λέει το κείμενο για τις απαιτήσει, θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα και τον Μάιο τουλάχιστον είχαμε αποτελέσματα για το ένα περιστατικό αλλά περιμένουμε και βάσει των πληροφοριών που πήραμε από την κυβέρνηση ότι και στις υπόλοιπες ε, περιπτώσεις θα έχουμε αποτελέσματα τουλάχιστον πρωτοβάθμια στην, ε, ε, στο μέλλον, άμεσα. Μόλις πάρουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία από το Κωσυφοπέδιο θα τα δώσουμε σε εσά στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Τάνια, θέλεις το λόγο? Ήθελα απλώς να ευχαριστήσω για την ε, πολύ αξιόλογη συνεισφορά των συναδέλφων και για τις πληροφορίες από την Κομισιόν. Θα ήθελα να συνεχίσει αυτό το θετικό πνεύμα στη συζήτηση. Θα δίνω σε εσάς ό,τι πληροφορία έχω. Ελπίζω ότι αυτά που απομένουν να γίνουν θα γίνουν πριν μπει σε ισχύ το καθεστώς ε, απελευθέρωσης. Είναι πάνω από 19 τα τεχνικά κριτήρια και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι όταν ε, πληρωθούν, εκπληρωθούν αυτά τα κριτήρια, δεν θα προσθέσουμε κάποιους όρους πολιτικούς. Η κάθε χώρα πρέπει να κρίνεται βάσει ε, της δικής της περίπτωσης. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, ότι ε, στην περίπτωση των συνόρων, ε, ας πούμε, πριν την κύρωση αυτή που απαιτείται, δεν, θα είχαμε, δεν το είχαμε το θέμα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα οδηγηθούμε στην κατάργηση των θεωρήσεων σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σήμερα. Η προθεσμία για την έκθεση φαγιών είναι 24 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι. Και τώρα θα ήθελα να σας πω πως το απόγευμα θα συνεχίσουμε με μία ακρόαση και επίσης με τα αποτελέσματα της ε, ε, αποστολής που πήγαμε στη Βιέννη. Οπότε θα μιλήσουμε και για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015. Σας ευχαριστώ πολύ.